Tutto pronto? Bene, eh, cari colleghi, eh, se volete... Καλώς αγαπητοί συνάδελφοι, αν την καλοσύνη καθίστε. Για να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας με κάποια λεπτά καθυστέρηση για να επιτρέψουμε και στους απόντες να καταφτάσουν εγκαίρως για την ψηφοφορία κάνουμε μια αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Το σημείο 7 που αφορά την έκθεση σχετικά με την αποστολή παρατήρησης εκλογών στο Κωσυφοπαίδιο θα εξεταστεί στην έκτακτη συνεδρίαση της επόμενης ε, Δευτέρας στο Στρασβούργο μετά από ανταλλαγή απόψεων με τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσης Σερβίας διέρισε Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις Θεωρώ ότι έχετε εγκρίνει την ημερήσια διάταξη με αυτή την ε, τροποποίηση που σας ανέφερα. Πρέπει να σας πω και άλλα πράγματα πριν ε, προβούμε στην προγραμματισμένη ψηφοφορία. Όπως γνωρίζετε το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια στην πρώτη ανάγνωση ενέκρινε την αναθεώρηση, την ομοθετική του μέσου για τη δημοκρατία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Συμβούλιο μετά ανακοίνωσε στο Κοινοβούλιο τη θέση του, την επίσημη, τον Δεκέμβριο. Τώρα θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία για τη δεύτερη ανάγνωση και η Επιτροπή μας θα πρέπει να καθορίσει τα ονόματα των δύο εισηγητών που θα έχουμε τις κυρίες Γκάλ και Λοκ Μπίλερ ως εισηγήτριες κατόπιν προτάσεως της ομάδας εργασίας όσον αφορά τις κατεξουδότηση πράξεις κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της για τα οικονομικά μέσα θα ψηφίσει το υιοθετημένο κείμενο με μεγάλη μάλλον υιοθέτηση στην πρώτη ανάγνωση το κείμενο. Θα ψηφίσει η Επιτροπή μας στις 26 Ιανουαρίου η στην Ολομέλη ψηφοφορία θα γίνει στην πρώτη σύνοδο του Φεβρουαρίου του 2010, λέει ο Πρόεδρος, 2011 και έτσι αρκετά γρήγορα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην προβλεπόμενη φάση της συνδιαλλαγής. Άρα δεν υπάρχουν δικές σας αντιρρήσεις. Δηλώνω επίσημα ότι οι συγγήτρες για τη δεύτερη ανάγνωση στον αυτό το θέμα αυτό είναι οι κυρίες Γκάλ και Λοκ Μπίλερ και η διαδικασία είναι η προβλεπόμενη και η αναφερόμενη. Επειδή βλέπω ότι είμαστε αρκετά πληροί στη σύνθεσή μας, μπορούμε να περάσουμε στη ψηφοφορία. Μπορείτε λοιπόν να εισαγάγετε την κάρτα σας στο ηλεκτρονικό μηχάνημα στη σχισμή ούτως ώστε να, να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία ηλεκτρονική. Μου αναφέρουν ότι ο κ. Κουμουτσάκος θέλει να πάρει το λόγο. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Ορίστε. Σας ακούμε κύριε Κουμουτσάκο. Σας ακούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εύχομαι καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους. Ε, θα ήθελα, πήρα, ζήτησα το λόγο για να αναφερθώ στο κείμενο στο οποίο πρόκειται να ψηφίσουμε για τη Frontex σε μια οριζόντια, οριζόντιου χαρακτήρα τροπολογία. Αφορά την χρήση του όρου παράνομος όταν χαρακτηρίζουμε την μετανάστευση ή παράτυπος illegal or irregular. Το κείμενο της Επιτροπής χρησιμοποιεί τον όρο illegal. Η αγαπητή εισηγήτρια προτείνει την αντεκατάστασή του με τον όρο irregular. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι το κείμενο που συζητάμε προσπαθεί να παντρέψει και να συνδυάσει την ανάγκη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας της Frontex και ταυτόχρονα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν πιστεύω ότι κανείς σε αυτή την αίθουσα είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το μονοπόλιο της ευαισθησίας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πόσο μάλλον το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και κύριε Πρόεδρε πρέπει να πω ότι πολλές φορές η κατάσταση στα σύνορα όταν αντιμετωπίζουμε αυτό το πολύ κρίσιμο φαινόμενο στα σύνορα της ελλάδας στον θαλάσσιο χώρο της μάλτας της ισπανίας ή της ιταλίας δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εμείς πιστεύουμε από τα γραφεία μας στις βρυξέλλες. η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη πολύ πιο κρίσιμη και πολύ πιο επικίνδυνη. γι' αυτό το λόγο προτείναμε να χρησιμοποιήσουμε να επιμείνουμε στον όρο illegal στο κείμενό μας και να μην συμφωνήσουμε με τον όρο irregular. σε μια προσπάθεια συμβιβασμού ανοιχτής διάθεσης και επικοδομητικής στάσης προτείνουμε και θα προτείνω να χρησιμοποιηθεί ο όρος clandestine ο οποίος κατά την άποψή μου είναι λιγότερο ισχυρός του illegal και σαφώς περισσότερο ισχυρός του irregular. Αυτό εναπόκειται στην ε, εισηγήτρια αν θέλει να το δεχθεί ως μια προσπάθεια συμβιβασμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, μπορούμε να ζητήσουμε από την, ε, τους τον εισηγητή, να μας πει. Κύριε Ροκμπίλερ, ποια είναι η απόψή της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρόταση. Δεν μπορώ όμως να τη δεχτώ. Θα παραμείνω με τη λέξη irregular. Ε, είναι κάτι συνηθισμένο που χρησιμοποιείται στη συζήτηση. Ακόμα και ο ίδιος ο επικεφαλής της Frontex χρησιμοποιεί τον όρο irregular Άρα δεν θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το, αυτή τη διατύπωση. Καλώς ο κ. Στάνοκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φοβάμαι παρόλο που βέβαια υποστηρίζω τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν θεωρώ ότι μετανάστευση ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν είναι δικαίωμα να μεταναστεύσει κανείς ε, στη χώρα μας. Και αν δεν έρθουν για νόμους λόγους και υποστούν κυρώσεις από τη χώρα υποδοχής ε, και δεν έχουν βάσιμο φόβο ε, για ότι διώκονται είναι παράνομη δικασία. Ίσως το clandestine να μην ακούγεται τόσο ε, δυνατό όσο το παράνομο όσο στα ελληνικά. στα αγγλικά σημαίνει σαν να είναι κάποιος παράνομος που είναι φυγόδικο και κρύβεται δικαιοσύνη. Το clandestine δεν ακούει τόσο καλά στα αγγλικά. Εγώ προτιμώ να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη illegal, να παραμείνουμε στη λέξη illegal αντί clandestine. Τελευταία παρέμβαση, όμως δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε συζήτηση από αυτού. Έχετε το λόγο. Κύριο Λούνατσεκ. Κυρία. Κυρία Λούνατσεκ. Για την ορολογία, ε, κύριε Τάνοκ, η διαδικασία μπορεί να είναι παράνομη, αλλά οι άνθρωποι δεν είναι παράνομοι, illegal. Και να επαναλάβω αυτό που είπε συνάδελφο. Αν ο επικεφαλή τη Frontex στα αγγλικά χρησιμοποιεί την ορολογία και λέει irregular, δεν νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κατέβει πιο κάτω από αυτό το όριο, να ξεφύγει από αυτό το πρότυπο. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Τροπολογία 2, στην οποία αναφερθήκατε, προτάθηκε από την εισηγήτρια με τον όρο irregular. Εάν δεν συμφωνείτε όσον αφορά αυτή την τροπολογία, εκείνος που είναι αντίθετος μπορεί να τοποθετηθεί κατά. Αν η συγγήτρια δεν συμφωνεί με την τροπολογία, υπάρχει δυνατότητα να ψηφίσει παραμένει άποψη, η προσέγγιση ε, ε, διαφορετική όπως είπε η συγγήτρια. Δεν μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή αν δεν συμφωνεί η συγγήτρια. Με αυτές τις διευκρινήσεις μπορούμε να προχωρήσουμε και να ψηφίσουμε που ξεκινάει η ψηφοφορία μας από τη συμβαστική 2 σε δύο τμήματα ξεχωριστά. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 5 που συμπεριλαμβάνει προφορική, ε, προφορική ψηφοφορία υπέρ, προφορική τροπολογία, συγγνώμη, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά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 Τροπολογία 7 κατά δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 7. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 22 κατά 19 υπέρ. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον απορρίπτεται, όμως δεν είμαι σίγουρος. Ας γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της συμβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Αυτή τη φορά εγκρίνεται 24 ψήφοι υπέρ, 19 κατά. Πάμε λοιπόν στην τροπολογία 41 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα ηλεκτρονικός έλεγχος όσον αφορά την τροπολογία 10 ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας ψηφοφορίας 24 ψήφοι αρνητικές, 21 θετικές, απορρίπτεται. Τροπολογία 45 με προφορική τροπολογία. Κύριε Κουμουτσάκο, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την ε, προφορική αυτή τροπολογία, υπάρχει μία πρόταση στην, ε, στην τροπολογία 45. Το κείμενο αναφέρεται σε applicable jurisdiction, maritime law provisions and relevant legislation. Προτείνω τη διαγραφή της αναφοράς maritime law provisions and έτσι το κείμενο μένει applicable jurisdiction and relevant legislation. Καλώς. Περιγράφει προφορική τροπολογία. Συμφωνώ. Μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν τη 45 με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία προφορική 11 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εγώ μάλλον νομίζω ότι απορρίπτεται αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από πλευρά παρισταμένων. Αυτό θεωρώ ότι συνέβη. Ας γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος, λοιπόν. Για το δεύτερο τμήμα της ε, τροπολογίας, προφορικής τροπολογίας 11, λέει ο Πρόεδρος. Ψηφίσατε όλοι. 26 όχι, 19 ναι, απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία την προφορική 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 52 αποσύρθηκε. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον εγκρίνεται. 57 έχει προφορική τροπολογία. Κύριε Κουμουτσάκο, θέλετε να μας παρουσιάσετε. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, η συγκεκριμένη τροπολογία ισχύει ακριβώς ό,τι ελέγχθη για την τροπολογία 45 η οποία ψηφίστηκε θετικά. Ευχαριστώ πολύ. Το, τον, τον jurisdiction. Είναι ακριβώς η ίδια με την πρότασή μου στο, στην τροπολογία 45 η οποία όπως σας είπα ψηφίστηκε από την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Καλώς. Δεν κατάλαβα γιατί δεν είχα διερμηνία. Όμως είναι πρακτικά ίδια. Α, ναι, ναι, ναι, το ακούω τώρα, ναι. Είναι η ίδια διευκρίνηση που κάνετε όπως αυτή που έγινε ήδη όσον αφορά τη 45. Ακολουθούμε τα ίδια κριτήρια, τσάγουμε τα ίδια κριτήρια. 57 λοιπόν με την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στη 12 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 58 είναι συμβατή. Την ψηφίζουμε λοιπόν. Υπέρ της 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Ζητείτε έλεγχος. Λοιπόν, για το πρώτο τμήμα της 13 ξεκινάει ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 20-25 εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 61 υπέρ, κατά. Δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα, οπότε γίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος όσον αφορά την τροπολογία 61. Ψήφισαν όλοι τώρα, πέρας ψηφοφόρειας. 26-21 απορρίπτεται. Τροπολογία 16 με προφορική τροπολογία. Παρέμβαση του κυρίου Κουμουτσάκου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είναι η τελευταία παρέμβαση που κάνω. Ε, στο σημείο αυτό υπάρχει μία αναφορά στην τροπολογία της εισηγήτριας η οποία λέει το εξής. With special regard to the right of everyone to leave a country including his or her own and international protection obligations with special regard to respect for the principle of non refoulement. Μπορούμε ε, να δεχθούμε το τμήμα, το πρώτο της προτάσεως της κυρίας Λογμπίλε, δηλαδή το κομμάτι που λέει «With special regard to the right of everyone to leave a country, including his or her own», αλλά όχι το υπόλοιπο τμήμα της τροπολογίας της. Εάν η κυρία Λογμπίλε ε, συμφωνεί, μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό. κυρία Λοκμπίλερ. Ευχαριστώ. Ναι, μπορώ να δεχτώ την πρόταση του κυρίου Κουμουτσάκου. Ε, Καλώς, λέει ο Πρόεδρος. Η εισηγήτρια δέχεται την πρότασή σας, οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε όπως ζητήσατε. Μία διευκρίνηση θα ήθελα όμως. Το δεύτερο τμήμα αφορά τη λέξη irregular αυτό είναι το δεύτερο τμήμα. Είναι κάτι άλλο. Άλλο σημείο που θέλετε να θίξετε σαν δεύτερο τμήμα. Είναι δικό μου το πρόβλημα, ίσως όχι δικό σας, αλλά δεν κατάλαβα ακριβώς ποιο είναι το δεύτερο τμήμα που θέλετε να θίξετε, να αναφέρετε. Κύριε Πρόεδρε, <clears throat> δεν είναι μόνο δικό σας πρόβλημα, είναι και δικό μου. Διότι αναφέρθηκα στην τροπολογία της κυρία Χλογμπίλα στο πρώτο κομμάτι που είναι, πρόκειται για δύο προτάσεις, μπορούμε να δεχτούμε την πρώτη αν πέσει η δεύτερη. Αν διαγράψουμε, τη δεύτερη, το δεύτερο τμήμα της προτάσεώς της. Αυτό το το είχαμε ξεχάσει. Το δεύτερο τμήμα ποιο είναι, αν έχετε την καλοσύνη να το διαβάσετε. Ε, η συγγήτριας έχει ως εξής with special regard to the right of everyone to leave a country including his or her own κομμάτι το οποίο μπορούμε να δεχτούμε και να μην δεχτούμε το δεύτερο τμήμα που είναι end international protection obligations with special regard to respect for the principle of non airful law. Καλώς. Τώρα είναι ξεκάθαρα. Ποιο είναι ξεκάθαρα το πρώτο και δεύτερο τμήμα. Αν δέχεται η συγγήτρια, η κυρία Λοκ Μπίλερ έχει το λόγο. Δέχεστε. Εντάξει, με αυτή τη διευκρίνηση ψηφίζουμε. Όσε τροποποιήθη λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 18, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64, υπέρ, κατά, δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος όσον αφορά την τροπολογία 64. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. 21 αρνητικές ψήφοι, 27 θετικές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 19 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική. Υπάρχει αίτημα ηλεκτρονικού ελέγχου όσον αφορά το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 19. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λείπουν δύο ψήφοι. Πέρας ψηφοφορίας. 25-22 απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές μάλλον απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 26 ξεκινάει η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας 19 κατά 25 υπέρ εγκρίνεται τροπολογία 2 Ορίστε. Κύριε Κουμουτσάκο, έχετε το λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, δεν τηρώ την υπόσχεσή μου να ήταν η τελευταία παρέμβασή μου προηγούμενη, γιατί μόλι τώρα ε, με ενημερώνουν ότι εδώ υπάρχει μια, ένα πρόβλημα στη λίστα του ΕΠΠ. Αντί για υπέρ είναι κατά στην τροπολογία που πρόκειται να ψηφίσουμε, την τροπολογία 2. Ευχαριστώ. Ναι, μετά αυτή τη διευκρίνηση που κάνατε στην αρχή, ναι, θα γίνει ιδιαίτερη διόρθωση. Λοιπόν, όσον αφορά το ΕΛΚ. Καλώς. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 α, ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινά ηλεκτρονικός έλεγχος όσον αφορά την τροπολογία 2 τέλος ψηφοφορίας Πέρα ψηφοφορία. 22 κατά, 26 υπέρ, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά. Δεν είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, ηλεκτρονικό έλεγχο όσον αφορά την 27. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 27. Τέλος. 29 κατά, 19 υπέρ, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 29. Ξεκινάει ψηφοφορία. 29. 29. Ξεκινάει η ψηφοφορια ψηφοφορία. Τέλος. 22-27 εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 32 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 32 ηλεκτρονικός έλεγχος που ξεκινάει ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας 23-26 εγκρίνεται. 34 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροποποιημένη πρόταση. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λείπει ένα συνάδελφος που δεν ψήφισε. Υπομονή όμως. Πέρας ψηφοφορία. 43 υπέρ, 5 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Εγκρίνεται το κείμενο. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε και να πάμε στη συζήτηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εμπορικές ε, προτιμήσεις κατεπίγουσες προτιμήσεις λοιπόν για το Πακιστάν. Είναι επιφορτισμένη η Επιτροπή μας με υποβολή γνωμοδότηση στην Επιτροπή ΙΝΤΑ. Η συγητής είναι ο κ. Πρέντα στον οποίο δίνω το λόγο για μια σύντομη παρέμβαση. Έχετε το λόγο, κύριε Πρέντα, όσον αφορά το θέμα που ε, είναι στη δική σας ευθύνη. Ευχαριστώ. Να περιμένω όμως λίγο να αποκατασταθεί κάποια ησυχία στην αίθουσα. Κύριε Πρόεδρε, δεν δούλεψε. Ψήφισα ναι, δεν δούλεψε το μηχάνημα. Τελική ψηφοφορία ψήφισα ναι. Εντάξει, το καταγράφουμε, λέει. Την ψήφο στη θετική, κύριε Μάουρο, όσον αφορά το προηγούμενο. Την ψηφοφορία που ήδη έχει ολοκληρωθεί. Διαλύεται το κοινό, αραιώνει. Θα σας, ακούμε πολύ καλά στα ακουστικά. Μπορείτε να, ακουσ, να ξεκινήσετε κύριε Πρέντα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το σχέδιο έκθεσης το σχέδιο μάλλον ε, κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει την παροχή αυτόνομων ε, τελωνιακών εμπορικών προτιμήσεων προς το Πακιστάν απαλλάσσοντας από υποχρέωση καταβολής φόρου 75 είδη προϊόντων που είναι ζωτική σημασία για τη χώρα αυτή, κυρίως ε, κλωστιφαντουργικά προϊόντα και προϊόντα ένδυσης. Η πρόταση αυτή Διακόπτει ο συγκεκριτής. Αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Μιλούμε και για ε, τις εμπορικές προτιμήσεις ό,τι αφορά την εθανόλη. Όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την οικονομική ανάκαμψη του Πακιστάν μετά τις ολέθρες ολέθριες πλημμύρες που έπλεξαν αυτή τη χώρα το καλοκαίρι του 2010 γιατί ο πληθυσμός στο λαό του Πακιστάν χρειάζεται την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και μια πιο μακροπρόθεσμη ενίσχυση ώστε να εξασφαλιστεί μια υφόρος ανάπτυξη για τη χώρα αυτή. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας παρέχει τη δυνατότητα να συνδυάσουμε αυτά τα δύο είδη δράσης, δηλαδή την ανθρωπιστική βοήθεια αφενός και την ε, υποστήριξη της αηφόρου ανάπτυξης αφετέρου. Τούτου λεχθέντος θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία που φαίνεται να δημιουργούν πρόβλημα στην πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και φαίνονται και από τις τροπολογίες που καταθέσαμε. Παρόλο που αυτές οι εμπορικές ε, προτιμήσεις θα έχουν τριετή διάρκεια, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν στηρίχθηκε σε εξαντλητική ανάλυση της επίπτωσης των μέτρων αυτών. Γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω περιορισμό αυτής της διάρκειας από την τριετία στη διετία, με δυνατότητα όμως παράταση κατά ένα ακόμη έτος, μετά από μια διεξοδική ανάλυση των επιπτώσεων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε και από τη σκοπιά το δικό μας ενδιαφερόντο ποια είναι η πραγματική επίπτωση των μέτρων αυτών στον πληθυσμό του Πακιστάν και να εξακριβώσουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των μέτρων και στους δημοσιονομικούς πόρους του Πακιστάν. Ιδιαίτερα μετά από την δέσμευση αυτής της χώρας να βελτιώσει το χρηματοπιστωτικό της σύστημα μετά από μία διετία θα μπορέσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει το πράσινο φως για την παράταση κατά ένα ακόμη έτος αυτών των ε, ε, προτιμήσεων. Αν γίνει φυσικά δεκτή αυτή η τροπολογία μου να περιοριστεί η διάρκεια σε μία διετία καταρχάς μέχρι ότου αναλυθούν διεξοδικά οι επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ κρίνω ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, μάλλον σε περίπτωση διαπίστωσης επιδείνωσης κατάστασης ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στο Πακιστάν θα ήταν αυτός από χρόνο λόγος για την αναστολή της συμφωνίας. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 18 Ιανουαρίου και ευχαριστώ. Λυπάμαι για αυτή τη δυσκολία, αλλά δυστυχώ είναι σχεδόν αναπόφευκτο όταν διεξάγεται μια ψηφοφορία να γίνεται κάποιο θόρυβο. Όμως τα ακουστικά ακούσαμε όλα όσα εσείς είχατε την καλοσύνη να παρουσιάσετε. Η κυρία Γκόμες έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον συνάδελφο Πρέντα για την εισαγωγή του θέματος που μας παρουσίασε και για την αιτιολόγησή του ως προς τις τροπολογίες που κατέθεσε. Συμφωνώ μαζί του ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συνάρτησή τους με την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί γνωρίζουμε από τις πακιστανικές αρχές ότι έχουν αναλάβει δέσμευση και θέλουν επέκταση αυτών των προτιμήσεων. Είναι εύκολο για την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δώσουν αυτές τις εμπορικές προτιμήσεις. Γιατί μιλούμε για κλωστιφαντουργία, δεν μιλούμε για αυτοκίνητα. Γι' αυτό είναι τόσο εύκολο και τόσο ελαφρά την καρδία δίνεται τις προτιμήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. μιλούσαμε για αυτοκίνητο βιομηχανία και τότε θα βλέπαμε πόσο εύκολη θα ήταν η παροχή τέτοιων προτιμήσεων αν ήταν περισσότεροι αυτοί που θα επηρεάζουν αυτά τα μέτρα, δεν ήταν η κλωστή φαντουργία που δεν είναι τόσο επίμαχο θέμα για το Συμβούλιο και την Επιτροπή, θα ήταν πολύ πιο επίμαχη η παροχή τέτοιων ε, προτιμήσεων. Πάντω, ε, ο τομέα αυτό όντω μπορεί να είναι τομέα ε, νευραλγικός για την οικονομική ανάπτυξη του Πακιστάν. Θα πρέπει όμω να εξασφαλίσουμε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η ανάπτυξη του κλωστή για την γενικότερη ανάκαμψη του Πακιστάν. Να προσέξουμε θέματα κοινωνικού ντάμπινγκ. Και μετά από τελευταία ανάλυση που έγινε, όπως μας υπενθύμησε και ο εισηγητής, δεν θα πρέπει να αμελούμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί εκεί υπάρχει πρόβλημα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα τα κάποια εργασιακά δικαιώματα που παραβιάζονται στο Πακιστάν. Συμφωνώ πάντως γενικά με τον εισηγητή και τονίζω και εγώ την ανάγκη να διενεργηθεί εξαντλητική διεξοδική μελέτη επιπτώσεων των μέτρων αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να κάνουμε παραχωρήσεις, να δίνουμε τέτοια αυτόνομα προνόμια χωρίς να πραγματοποιούμε προηγουμένως μια διεξοδική ανάλυση των επιπτώσεών τους. Άλλωστε και στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου δεν θα είναι εύκολο να περάσουν κατά τέτοια μέτρα, γιατί και άλλε χώρε τη περιοχή αυτή που είναι παραγωγή έχουν αμφιβολίε ω προ την επέκταση αυτών των προνομίων. Και ε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να δείξουμε την αλληλεγγύη μα προ το Πακιστάν. Και ίσω οι άλλοι αυτοί τρόποι μπορεί να είναι και πιο χρήσιμοι για την βιομηχανική ανάπτυξη του Πακιστάν. και φυσικά με απόλυτο σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα είμαι όμως αρνητική. Είναι σημαντικό στις, στη γνωμοδότησή μας να εκφράσουμε τις επιφυλάξεις μας που είναι σοβαρές και νομίζω ότι αυτό γίνεται δεόντως από τον εισηγητή μας. Πάντως μέχρι τις 18 Ιανουαρίου, παρόλο που είναι σύντομη προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών, θα συμβάλλω και εγώ με δικές μου τροπολογίες. Καλώς, δεν ζήτησε άλλο το λόγο. Οπότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος. Η Επιτροπή σχεδία σε την ε, υιοθέτηση του θέματος 26 Ιανουαρίου, οπότε η προθεσμία είναι πολύ περιορισμένη. Οι τροπολογίες μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 18 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι και η ψηφοφορία στην Επιτροπή προβλέπεται στις 25 Ιανουαρίου. Είναι τόσο περιορισμένο το χρονικό διάστημα και γι' αυτό σας συμβουλεύουμε, μάλλον προτείνουμε στους συναδέλφους να υποβάλουν στα αγγλικά τις τροπολογίες. Πάμε τώρα στο σχέδιο έκθεσης και τις σχετικές τροπολογίες. των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με το Ιράν. Η συγγητής είναι ο κύριος Μπέλτερ, ο οποίος έχει το λόγο. Σας ακούμε, κύριε Μπέλτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για τις τροπολογίες που καταθέσατε και δείχνουν το ενδιαφέρον σας στην σημαντική αυτή έκθεση και η πρόθεσή μου είναι να καταλήξουμε βεβαίω σε μια επικοδομητική κυβέρνηση για να εξυπηρετεί βεβαίω και τον δυναμικό και ταλαντούχο λαό του Ιράν. Βεβαίω, αυτή τη στιγμή διεθνώ ξεκινάει, ξεκίνησε τον πρώτο μήνα ο πρώτο γύρος διαπραγματεύσεων στην Γενέβη και αυτό το μήνα ερχόμαστε ε, σε επίκαιρη στιγμή με μια στιβαρή έκθεση θα έλεγα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αυτά ως βάση είδα όλες τις ε, τροπολογίες της ζήγησα θα έλεγα και θα σας πω τώρα τις πρώτες μου σκέψεις για τις τροπολογίες αυτές. και βεβαίως είδα πάρα πολλές ε, τροπολογίες ε, που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελπίζω να μπορέσουν να συμβαστούν να συνενωθούν σε κάποιες συμβαστικές ε, τροπολογίες. Ούτως ή άλλως ε, οι προθεσμίες ήταν πάρα πολύ σύντομες και ελπίζω να έχουμε αυτή την εβδομάδα ή την ερχόμενη εβδομάδα τις αντιδράσεις σας και έτσι είτε διμερός είτε όλοι μαζί να μπορέσουμε να συζητήσουμε την αντιμετώπιση μας. Έχοντας πει αυτά, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, να αναφερθώ λίγο σε ποιες τροπολογίες μπορώ να στηρίξω αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή το τονίζω αυτό. Γιατί, όπως είπα, αξίζουν όλες ε, να εξεταστούν λεπτομερέστερα. Λοιπόν, όσον αφορά τα εκτιμώντας α, εγώ θα πρότεινα να μείνει το κείμενο ως έχει. Στο β, τροπολογία είναι κάποια βελτίωση. Στο σε έχουμε την 43 και 44. Στο Δέλτα. Νομίζω μπορούμε να, να δούμε τροπολογία της κυρίας ε, Γκόμες. Είναι αρκετά επικοδομητική. Θα ήθελα να τη δούμε οι δυο μας. Ή για την 48 είναι μια βελτίωση. Η F ε, προσπάθησα να κάνω μια, ένα συμβιβασμό. Ε, κατέθεσα κάποιες ε, προτάσεις στους σκιώδεις εισηγητές για τις 52 ε, και 53 μετά στο C και το G δυστυχώς εδώ πέρα δεν μπορώ να συμφωνήσω νομίζω πως ε, θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη για τη θέση της Τουρκίας όσον αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ιράν. Όπως είπα αυτή τη στιγμή δεν νομίζω να μπορώ να το δεχτώ μετά στις παραγράφους. Στην 1 για την 76 πράγματι μπορώ να τη ρίξω. Στη 2 δηλαδή η τροπολογία 81 είναι βελτίωση. Στην 3 θέλω να μείνει όπως είναι. 4 η 101 είναι βελτίωση. Στην 5 θέλω να μείνει όπως είναι. 6 νομίζω εκεί πέρα δεν έχει υποβληθεί κάτι. Στην 7 130 και 135 νομίζω μπορούμε να βρούμε ένα συμβασμό. 8 επίσης αναγκαία συμπλήρωση. 9 για 157, 58, 59 δεν είναι τόσο συμβαστικές οι τροπολογίες. Νομίζω έχουν κατατεθεί τρεις φορές το, το ίδιο πράγμα και εδώ πέρα νομίζω μειώνεται και η σημασία τους. Για το 9 σας είπα λοιπόν ότι είναι ταυτόσιμες, ε, μπορώ να τις στηρίξω. Στην 10 Εδώ πέρα μπορώ να δεχτώ την 164, αλλά πρέπει να συγκριθεί και με άλλε. Στην 11 συμφωνώ με την 166, 167, 168. Στη 12 πρέπει να πω πως αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να συμφωνήσω με τις τροπολογίες που προτείνονται. Στην παράγραφο 13 ισχύει αυτό το οποίο είπε για την 179, 180, 181. Δηλαδή μπορώ να στηρίξω την 181 και μετά υπάρχει μια σειρά συμβαστικών παραγράφων. Στην 15 ε, από αποπειράθηκα να κάνω έναν συμβιβασμό. με βάση την 193 μέχρι 197 και την 208-209, ε, μετά η συμβα... συμβαστική 17 συμπεριλαμβάνει την 225 και 223, στην 18 δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάποιον συμβασμό, 19 συμβασμός ε, από την 242 μέχρι 244, με την 20 την 55, 56, 57 21 όχι, 22 ξανά επανέρχεται η Τουρκία και στην 23 έχουμε την 298 η οποία είναι ταυτόσιμη οπότε νομίζω δεν χρειάζεται και μετά έχουμε μια συμβαστική λύση για την θανατική ποινή ελπίζω εδώ πέρα τις επόμενες ημέρες να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και με τους και τέλος μπορώ να στηρίξω τις εξής τροπολογίες 1, 4, 5, 6, 8, 9, 30, 43, 90, 93, 44, 110, Επίσης αυτό το οποίο αναφέρεται για την ε, Μπαϊράμι που έχει καταδικαστεί σε θάνατο για αυτή την ε, Ιρανή ορολανδικής καταγωγής 138, 139, 141, 47 185, 186, 200, 201, 202, 203, 204, 213, 215, 219 να την συζητήσουμε, 226, 238, 266, 265, 283, 284 και τέλος 301. Ευχαριστώ συνάδελφοι, ελπίζω με την ίδια επιμέλεια να παρακολουθήσουμε το θέμα. Είμαι πάντα βέβαιος στη διάθεσή σας για επαφές και βεβαίως προβλέπεται η ψηφοφορία για την 1η Φεβρουαρίου οπότε υπάρχει ακόμα λίγος χρόνος αλλά βεβαίως κάνει πιο περίπλοκη την κατάσταση πως καμιά φορά έχουν κατατεθεί τροπολογίες οι οποίες πηγαίνουν σε αντίθετες ε, κατευθύνσεις οπότε προσπαθούμε να κάνουμε μια αρκετά δυνατή έκθεση θα έλεγα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την συνεργασία σας και τα σχόλιά σας και έχουμε ακόμα κάποιες εβδομάδες οι οποίες ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Μπέλντερ. Το λόγο τον έχει κυρία Μούνιτς. Ε, ευχαριστώ. Για την έκθεση αυτή έχουν κατατεθεί 300 τροπολογίε ε, που δείχνουν το ζωηρό ενδιαφέρον που προκάλεσε, όπω είπε και ο κ. Μπέλντερ. 300 τροπολογίε κατατέθηκαν γιατί δεν υπήρχε συμφωνία προ τη βάση που υιοθέτησε ο εισηγητή Μπέλντερ. Και Πολλές από τις τροπολογίες αυτές είτε είναι πανομοιότυπες είτε είναι κοινέ μεταξύ των πολιτικών ομάδων και μάλιστα πολιτικών ομάδων που γενικώ δεν συμφωνούν στις θέσεις τους. Αυτό νομίζω θα πρέπει να προβληματίσει τον κύριο Μπέλντερ για την έκθεση που μας υπέβαλε για το έγγραφο εργασία του. Ευχαριστώ για τις συμβαστικές τροπολογίες που καταθέσατε. Θα είναι η βάση για περαιτέρω επεξεργασία, αλλά λυπούμε που δεν έγινε καμία συνεδρίαση με τους σκιώδεις ηγητές, γιατί πραγματικά η έκθεση είναι πολύ περίπλοκη, το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο, η θέση της, της χώρας αυτής στην περιοχή είναι πολύ στρατηγική και έχει σχέση και η θέση της στα Ηνωμένα Έθνη και η διμερή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα όπως είναι τα πυρηνικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αστάθεια στην περιοχή, η σχέση με το Αφγανιστάν, οι επιπτώσεις ε, για το Αφγανιστάν. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα και θα έπρεπε να είχατε επιδιώξει μια μεγαλύτερη συνένεση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κάτι που δεν συνέβη, όπως φάνηκε από την έλλειψη συνεννοήσεων και συνεδριάσεων με τους κοιόδης ηγητές. Θα αναλύσουμε τις ε, συμβαστικές αστροπολογίες πάντως και θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Σε ό,τι αφορά την αιτιολογική σκέψη F, διαφωνούμε με την ε, δερμία φρασεολογία που χρησιμοποιείται για την έννοια της απειλής στην ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής. Εμείς προτιμούμε τη διατύπωση των τροπολογιών 48, 49 και 50 Τρει τροπολογίες από διαφορετικές πολιτικές ομάδες προτείνουν κάτι τελείω διαφορετικό κύριε Μπέλντερ και υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η ρευστότητα των σχέσεων του Ιράν με τις γειτονικέ χώρες και όχι ο σταθεροποιητικό χαρακτήρα του Ιράν για την περιοχή. Άλλη είναι η καλύτερη διατύπωση, λιγότερο οξύ από τη δική σα. Επίση, ε, η επιθετική αυτή φρασιολογία ε, κατά του Ισραήλ και η υποστήριξη της Χαμάς και του Χεσπολάχ είναι θέμα πολύ πιο ανησυχητικά. Αυτά θα πρέπει να τα διατηρήσουμε στην έκθεση. Αλλά προσοχή στην φρασολογία για την σχέση του Ιράν με τις γειτονικέ χώρες. Σε ό,τι αφορά τη συμβαστική τροπολογία 3, νομίζω ότι θα πρέπει ρητά να αναφερθούν οι προσπάθειες του Ιράν για τις παρεμβάσεις στο ίντερνετ ε, ε, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, όπω αναφέρει η τροπολογία 142 του κ. Τάνοκ. Επίση, για την αξιοπιστή της έκθεσης θα πρέπει να αναφέρουμε και τα μέσα ε, ε, μαζική ενημέρωσης ή τα, ευρωπαϊκέ τις ευρωπαϊκές εφημερίδες, των οποίων οι ειδικοί επισταλμένοι απελάθηκαν από το Ιράν, όπως είναι οι δημοσιογράφοι της ΠαΐΣ και του Guardian για την παράγραφο 17 δεν μπορούμε να περιοριστούμε μόνο στο διάλογο και τις συζητήσεις που έγιναν με το Ιράν. Νομίζω θα μπορούσαμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι, πιο διορατικοί και να λάβουμε υπόψη και τις συνομιλίες ε, στη Γενέβη. το, ε, το 5 συν 1 και τις ε, επικείμενες ε, συζητήσεις της 25ης Ιανουαρίου στην Κωνσταντινούπολη. Και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε εκτό από τα πυρηνικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για άλλου τομεί σχέσεων με το Ιράν, Όπω είναι η εσωτερική πολιτική και η περιφερειακή ασφάλεια. Νομίζω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε την παράγραφο αυτή για να διευρύνουμε κάπως το περιεχόμενό τη και να μην περιοριστούμε μόνο στα πυρηνικά. Σε ό,τι αφορά τη συμβαστική τροπολογία 7 για την παράγραφο 20, νομίζω ότι θα ήταν εσφαλμένο να μην γίνει καμία διαφοροποίηση μεταξύ των ποιον στις ε, Ιρανικές αρχές ή στην Ιρανική ηγεσία συνιστούν μια απειλή ή ε, εκφράστηκαν απειλητικά εις βάρος του Ισραήλ. Γιατί οι δηλώσεις αυτές έγιναν κυρίως από τον Αχματινετζάντ. Όχι από την Ιρανική ηγεσία γενικώ. Θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση και να δούμε ποιο ακριβώ έκανε αυτέ τι δηλώσει για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε, να διατηρήσουμε επικοινωνίας και τον πολιτικό διάλογο με το Ιράν. Να κάνουμε διάκριση το ποιο έκανε τι δηλώσει αυτέ στο Ιράν και να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Γιατί υπάρχουν πολιτικέ δυνάμει στο Ιράν με τι οποίε μπορούμε να έχουμε μια βάση επικοινωνία και ένα διάλογο. Αυτά ω προ τι συμβαστικέ λύσει. Για τι υπόλοιπε που δεν ανέφερα δεν έχουμε πρόβλημα. Και νομίζω ότι επήγει μια συνεδρίαση με τους σκιώδεις συγητές. Θα πρέπει να καταλήξουμε στις συμβαστικές λύσεις και για τις πιο επίμαχες τροπολογίες. Και σε περίπτωση που δεν καταλήξουμε συμφωνία μεταξύ των σκιωδών εισηγητών και του εισηγητού, θα πρέπει να ψηφίσουμε κάθε τροπολογία ξεχωριστά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Μούνιθ. Η κυρία Λόκμπιλερ έχει το λόγο. Πρόεδρος Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Ιράν. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στι συζητήσεις για αυτά τα οποία προτείνει ο κύριος Μπέλντερ εδώ πέρα. Νομίζω πως συνεννοηθήκαμε πως πρέπει να έχει τρεις βασικές γραμμές η έκθεση. Σε εσωτερικές εξελίξεις, ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατικές εξελίξεις και την οικονομική ανάπτυξη. Και μετά ο πυρηνικός φάκελος και τρίτον ο ρόλος του Ιράν στην περιοχή. Και τρεις αυτοί τομείς νομίζω θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με βάση την πολιτική double track, δηλαδή να αποφευχθούν οι παρανοήσεις, να ασκήσουμε πίεση και να δείξουμε πως είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω πως η πρόταση δεν ε, επαρκούσε, δεν έφτανε σε αυτό το επίπεδο την προηγούμενη φορά. Και τώρα έχουμε 298 τροπολογίες. Πράγματι είναι τιτάνιο αυτό το έργο, αλλά δεν είναι επιφανειακές και με πολεμική διάθεση. Είναι ουσιαστικές αυτές οι τροπολογίες, εξειδικεύουν απαιτήσει, συνδέουν το πώς μπορεί να συνεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλους πολυμερείς οργανισμούς και εν μέρη αυτές οι τροπολογίες είναι, έχουν συνοψιστεί. Π.χ. η ομάδα μου, η πράσινη, συνεργάστηκε πάρα πολύ με τους σοσιαλιστές ήμασταν πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Με αυτές λοιπόν τις οχτώ συμβαστικές ε, τροπολογίες που ε, είδαμε χτες, μιλάμε για 34 ε, τροπολογίες ε, οι οποίες συμβάζονται εδώ πέρα. Τα είπατε πάρα πολύ γρήγορα κάποιες τροπολογίες τις οποίες δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω. Νομίζω πως ε, εδώ πέρα ε, δεν είναι σωστή αυτή η αντιμετώπιση γιατί όλες αυτές οι συμβαστικές τροπολογίες αφο... έφυγαν στις συμβαστικές τροπολογίες όλα όσα αφορούν τον περιφερειακό ρόλο του Ιράν στην περιοχή. Οπότε θα πρέπει νομίζω να δούμε τα πράγματα και συζητώντας Πράγματι προσφέρατε διμερείς επαφές, πράγματι έτσι θα πρέπει να συνεννοηθούμε, αλλά χρειάζεται χρόνος και να προετοιμαστούμε καλύτερα και να συναντηθούμε ισχυώδεις. Γιατί η έκθεση αυτή πρέπει να αποτελέσει την βάση για την περαιτέρω πολιτική, ε, την Ιρανική του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Λόκ Μπίλερ. Ο κ. μου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Μπέλτερ, όντως αν έχουν κατατεθεί τόσες πολλές τροπολογίες, είναι ότι είναι συναρπαστικό το θέμα. Αλλά να μιλήσουμε για πάθος, ότι μας έχει παθιάσει το θέμα γιατί το Ιράν, νομίζω ότι είναι άκερη και αδόκιμη κρίση. Σίγουρα το Ιράν έχει στρατηγική θέση για το σύνολο της παγκόσμιας κοινότητας και έχουμε καταθέσει τόσες τροπολογίες γιατί ανησυχούμε ότι δεν θα σταθεί στο ύψο των περιστάσεων αυτή η έκθεση και δεν θα συμβάλλει στην απεμπλοκή της ανησυχητικής αυτής κατάστασης. Πολύ συχνά λέμε ότι ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με αγαθές προθέσεις. Προσοχή λοιπόν, γιατί μερικές φορές οι αγαθές προθέσεις δεν καταλήγουν σε καλά αποτελέσματα. Και το γεγονός ότι θέλετε να επικεντρώσετε έκθεση, την έκθεση σε ένα συγκεκριμένο θέμα και αρκετά μανιχαριστικό τρόπο, αυτό θα μας οδηγήσει σε μία αποδυνάμωση. Δεν θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε την απαραίτητη συνένεση, την ομοφωνία που χρειάζεται ουσιαστικά για να αποκτήσει αυτή η έκθεση μια πολιτική ισχύ και να διατρανώσει τη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να γίνει αυτή η ακουστεί. Δεν είμαι ή εισηγητής, αλλά ε, δεν φαίνεται ότι έχετε συνεννοηθεί με τους σκιώδης ηγητές για να καταλήξετε τι συμβαστικές λύσεις που θα γίνουν κοινώς αποδεκτές. Δεν θα πρέπει να φανεί στο θέμα αυτό είμαστε διχασμένοι, γιατί έτσι θα βάλουμε το κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μια τέτοια διαφωνία μεταξύ μας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη κάποιες τροπολογίες, κύριε Σιγητά, γιατί επισημάναμε αρκετά προβληματικά σημεία στην έκθεση. Καταρχήν θα πρέπει να έρθει οποιαδήποτε αφησημία στο κείμενο σε ό,τι αφορά το, τη σύγκρουση των πολιτισμών, όπως λέγαμε παλιά. Γιατί αυτό πραγματικά θα παίξει το παιχνίδι των Ιρανών φονταμενταλιστών. Γιατί, όπως ξέρετε, η σύγκρουση δεν γίνεται μεταξύ Δύση και Ιράν. Γιατί και πολλές μουσουλμανικές και αραβικές γειτονικές χώρες δεν υποστηρίζουν αυτή τη θέση. Αν μείνουμε λοιπόν σε αυτή την μανιχαριστική προσέγγιση θα διαπράξουμε ένα κολοσιαίο λάθος. Και γι' αυτό καταθέσαμε τροπολογίες για να τροποποιήσουμε αυτή τη διατύπωση. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο σημείο αυτό. Επίσης να μην κάνουμε λάθος και ως προς την ιστορία του Ιράν. Το θέμα των πυρηνικών ε, είτε, με, είτε στρατιωτικού, για στρατιωτικούς σκοπούς είτε μη στρατιωτικούς δεν σχετίζεται μόνο με το τωρινό καθεστώς. Υπάρχει μια ιστορία στο Ιράν. Υπάρχει η δηλωμένη βούληση του Ιράν να κτίσει μια θέση που έχει στην ιστορία. Δεν είναι μόνο αυτό το καθεστώς που ασχολείται με τα πυρηνικά και αυτό το θέμα θα συνεχιστεί και αργότερα. Και αυτό αλλάζει τον τρόπο προσέγγισης, ε, το δικό μας ως προς τα θέματα αυτά. Θα πρέπει να το δούμε και από ιστορική σκοπιά. Αναφέρεστε σε μια ιδεολογία, αλλά δεν φαίνεται να τη τηρείτε. Υπάρχει περίφημη διπλή προσέγγιση της κύρωσης αφενός και της ε, διαπραγμάτευση αφετέρου. Στο κείμενο όμως που μας υποβάλλεται σήμερα, παρόλο που επανεπιβεβαιώνεται αυτή την ανάγκη της διπλής προσέγγισης, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια ανισορροπία στην έκθεσή σας. Δεν βλέπουμε εμείς καμία θετική προοπτική. Πώς ε, θα μπορέσουμε να έχουμε διάλογο με την κοινωνία των πολιτών στο Ιράν και να την παροτρύνουμε και την πολιτική ε, ηγεσία για μια πρόοδο. Και νομίζω ότι και με τις αμερικανικές προσπάθειες και τις, ε, την πολιτική του Ομπάμα και την ε, έμφαση που δόθηκε στο διάλογο και τη δυνατότητα επανένταξης του Ιράν στην παγκόσμια κοινότητα, σε αυτά τα θέματα θα πρέπει και εμείς ε, να επικεντρωθούμε και να μην εστιαστούμε μόνο στο θέμα των κυρώσεων. Θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την ισορροπία του κειμένου προς τη διπλή προσέγγιση. Επειδή είμαστε υπέρ του θέματος και των κυρώσεων, καλό θα ήταν να κάνουμε μια πιο διεξοδική ανάλυση και πιο εμπεριστατωμένη, όπως μας υπενθύμησε η πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Ιράν. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πιο εμπεριστατωμένη και πιο ακριβή η ανάλυση της έκθεσης για την πραγματικότητα της κοινωνίας του Ιράν. Όχι μόνο πέντε παράγραφοι δηλαδή, εκ των οποίων οι δύο αναφέρονται στους Ισλαμ, στους ε, φρουρούς της Επανάστασης, στο σώμα των Ισλαμικών φρουρών της Επανάστασης. Επίσης θα πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματική πολιτικότητα των κυρώσεων, η πολιτική πραγματικότητα των κυρώσεων και ποιες ε, είναι οι αναμενόμενες συνέπειες και για την Ιρανική κοινωνία. Νομίζω ότι με μια ακριβέστερη προσέγγιση θα είμαστε και εμείς αφέστεροι απέναντι στην Ιρανική κοινωνία που ουσιαστικά είναι αυτή που θέλουμε να υποστηρίξουμε. Δεν θα επισέλθω τώρα σε λεπτομέρειες των τροπολογιών. Δεν ε, μελέτησα ακόμη διεξοδικά ε, τις ε, συμβαστικές σας τροπολογίες. Είδα το κατάλογο ψηφοφορίας σας, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστός αυτός ο τρόπος για να επιδιώξουμε τη συνένεση. Σημερίζομαι τις ανησυχίες σας, αλλά στόχος είναι να είμαστε αποτελεσματικοί. Θα πρέπει να επιδιώξετε μία συνένεση. Νομίζω ότι αυτό είναι ο πιο υπεύθυνο τρόπος ε, και καλύτερη μεθοδολογία. Σας ευχαριστώ κύριε Πεγιόν. Ο κύριος Γκάλερ έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Μπέλτερ για τις συμβαστικές τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και για τις εξηγήσεις του. για το πώς βλέπει τις διάφορες τροπολογίες. Και εγώ θεωρώ πρώτα απ' όλα πως πράγματι πρέπει να συναντηθούμε οι σκιώδεις και στο πλαίσιο αυτό νομίζω τους μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κοινή ευρύτερη ε, προσέγγιση και στάση άρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εναντί του Ιράν. Είναι πολιτικά σημαντικό όχι μόνο το Κοινοβούλιο, αλλά συνολικά η διεθνής κοινότητα και οπωσδήποτε ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει μία κοινή στάση εναντί του καθεστώτος εκεί πέρα. Θεωρώ πως ε, για το χαρακτήρα του καθεστώτος δεν υπάρχει καμία διαφωνία σοβαρή και το αποτέλεσμα βεβαίως είναι πως ε, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την περιγραφή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια συνένεση στην περιγραφή αλλά και στις λεπτομέρειες μετά όσον αφορά τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουμε για να βοηθήσουμε την Ιρανική κοινωνία των πολιτών στον αγώνα της για περισσότερη δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Εκεί πέρα ε, νομίζω υπάρχει αρκετά μεγάλη δυνατότητα συμβασμού. Όσον αφορά το πυρηνικό ζήτημα, εξακολουθούμε νομίζω. Ευτυχώς και εδώ πέρα να έχουμε μια κοινή στάση έναντι του Ιράν. Οπωσδήποτε βεβαίως Ευρωπαίοι και Αμερικανοί θα ήθελαν να πάνε λίγο παραπέρα όσον αφορά τις κυρώσεις. Η στάση της ομάδας μας είναι ξεκάθαρη. Δηλαδή θα πρέπει να ζητήσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια αυτό το οποίο ζητάει δηλαδή και η Διεθνής Υπηρεσία Τοπικής Ενέργειας, πλήρη συνεργασία. Το θέμα αυτό νομίζω μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα κείμενο το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο συνένεσης, όπως και σε προηγούμενα ε, ψηφίσματα. Όσον αφορά τώρα την εκτίμηση του Ιράν ε, και του ρόλου του στην περιοχή. Εκεί πέρα διαπιστώνουμε πως ε, υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις, αλλά εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θεωρούμε πως ε, το Ιράν αποτελεί κίνδυνο για την περιοχή, όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά και για άλλους γείτονες. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει πως θα αναστείλουμε το διάλογο και τις επαφές. Αντιθέτως, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν για να ξεκαθαρίσουμε στους κρατούντες το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Κάτι το πιο συγκεκριμένο τώρα όσον αφορά την εκτίμηση του ρόλου της Τουρκίας. Εκεί ε, δεν θα ήθελα εγώ να πω πως έχει κάποια άλλα κίνητρα η Τουρκία με τις επαφές της με το Ιράν αλλά πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα αυτό με την Τουρκία να έχουμε διάλογο μεταξύ της νομίζω πως η Τουρκία μπορεί να επιδείξει επικοδομητικό ρόλο οπότε εγώ δεν θα ήθελα να πω τίποτα το αρνητικό όσον αφορά αυτές τις επαφές. Θεωρώ επίσης πως πρέπει στην έκθεση να δούμε πού υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Αυτό, παραδείγματος χάρη, είναι στην... Αυτό στοχεύει και η τροπολογία Μπροκ ότι δηλαδή θα πρέπει να συμμετάσχει προσεχώς σε μια θετική εξέλιξη στο Αφγανιστάν το Ιράν ε, δηλαδή όσον αφορά την καταπολέμηση του εμπορίου των ναρκωτικών όπου έχουμε να συμφέροντα και μπορούμε να, να συνεργαστούμε με το Ιράν και αυτή η πτυχή νομίζω πρέπει να αποσαφινιστεί. Θεωρώ λοιπόν πως ε, θα καταλήξουμε με τον εισηγητή σε μια καλή έκθεση και το χαρτί που έχουμε μπροστά μας είναι μια καλή βάση νομίζω. Όλα τα υπόλοιπα θα λυθούν σε συναντήσεις με τους κοιόδης εισηγητές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σάκη, επόμενος ομιλητής. Κυρία Σάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή τον κύριο Μπέλτερ και τους συναδέλφους. Αναφέρθηκαν πολλά και υπάρχει διάθεση επικοδομητικής συνεργασίας. Προσβλέπουμε σε αυτό. Ε, θέλω κάποιες διευκρινήσεις. Παρόλο που η συγητής μιλάει τη μητρική μου γλώσσα και σημείωνα όσο πιο γρήγορα μπορούσα, μου ξέφυγαν κάποιες λεπτομέρειες και θέλω κάποιες διευκρινήσεις για τα εξής. Ο εισηγητής αναφερόταν στις συμβαστικές τροπολογίες και θεώρησε ότι είπε ότι επειδή υπήρχαν πολλές τροπολογίες που υπευλήθησαν, που ήταν ταυτόσιμες, ότι αυτός δεν είναι λόγος για να σχηματίσουν συμβαστική τροπολογία. Εγώ πιστεύω ότι το ότι κάποιες ομάδες υπέβαλαν τις τροπολογίες, αυτό δείχνει ότι υπάρχει κοινή αίσθηση ότι έχουν σημασία οι τροπολογίε. Οπότε θα ήταν πολύ καλό να υπάρξει μια, δημιουργηθεί μια βάση για συμβαστική τροπολογία. Άλλο ερώτημα γενική φύσεω. Θα είμαστε συγκεκριμένοι για κάποιε περιπτώσει ή θέλουμε να εστιαστούμε σε κάποιε από τι βασικέ ανησυχίε πιο γενικόλογα. Αυτό ισχύει για την κατονομασία συγκεκριμένων ε, υποθέσεων όσον αφορά την ε, θανατική ποινή που εφαρμόζεται σε πρώτερες Εκθέσει ήταν βασικό θέμα. Θα αναφέραμε συγκεκριμένε υποθέσεις, περιπτώσεις ή όχι. Πια είναι η άποψη του εισηγητή. Για να είμαστε επικοδομητικοί, κάτι που όλοι επιθυμούμε, η ε, διατύπωση, ο τρόπο που διατυπώνουμε την άποψή μα για το Ιράν είναι σημαντικότατη. Θέλουμε να αντικατοπτρίζονται οι ανησυχίε όποιο αντικειμενικά γίνεται. Οι ανησυχίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήταν καλό αν το πετυχαίναμε αυτό. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην Τουρκία και ο συγητής αναφέρθηκε στι αποκλίνουσε απόψει στον αφορά το θέμα. Παρακαλώ του συναδέλφου να μην χρησιμοποιούν αυτή την έκθεση για να εκφράζουν γενική στάση στον αφορά την Τουρκία, αλλά να δούμε τρόπου με τον οποίο ε, θα μπορεί η Τουρκία να είναι πιο επικοδομητική έναντι του Ιράν. Σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να διευκρινιστεί διατύπωση. Σίγουρα θα τα καταφέρουμε αυτά όταν συναντηθούμε τους κοιόδης. Δεν θα επιστρέψω αυτό το, στις Γενικώ πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντικό να είμαστε όσο το πιο δυνατόν συγκεκριμένοι να κάνουμε διάκριση μεταξύ του λαού του Ιράν και της κυβερνήσεως της χώρας αυτής. Θέλουμε να προσελκύσουμε, να δημιουργήσουμε υποστήριξη, να στηρίξουμε το λαό του Ιράν στις ειρηνικέ του διεκδικήσεις για περισσότερε ελευθερίες και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και Θέλουμε το καθεστώς να σέβεται ανθρώπινα δικαιώματα. Όσον αφορά τι ευθύνε. Έχει ευθύνε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια κράτη-μέλη έχουν δεχτεί πρόσφυγες από το Ιράν. Και χαίρομαι που η συγητής είναι πρόθυμος να υποστηρίξει τη σχετική τροπολογία που αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση αυτό είπε. Ποια είναι η άποψη του συγητού μετά για τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων για άτομα της κυβερνήσεως, για ε, άτομα, για υπεύθυνους της κυβερνήσεως ε, του Ιράν που είναι υπεύθυνα που είναι υπεύθυνοι μάλλον για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Περιμένω τις διευκρινήσεις, προσβλέπω συνεργασία με όλους τους συναδέλφους για να έχουμε μια πιο επικοδομητική έκθεση, πιο περιεκτική έκθεση για αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να προσπαθήσουμε τόσο ώστε να συνεργαστούμε όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Σάκε. Λέζινγκ. Η κυρία Λέζινγκ είναι η επόμενη αγορήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μπέλντερ. Δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες όσον αφορά την κάθε τροπολογία. Θα αναφερθώ στις βασικές γραμμές ε, της Τοποθέτηση τη ομάδα μου. Και στην τελευταία συνάντησή μας το είχα πει και εδώ πέρα θέλω να επαναλάβω την δύσκολη πολιτική και οικονομική κατάσταση και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, τα οποία δεν τα αρνούμε, δεν τα αρνούμε. Αλλά πρέπει να πω πως η ομάδα μου και εγώ ασκούμε κριτική σε αυτή την έκθεση και δεν θα μπορέσουμε να την υπερψηφίσουμε. Εμείς είμαστε υπέρ μιας στρατηγικής αλλαγής και αλλαγής πολιτικής της Ένωσης και των ΗΠΑ με στόχο να σπάσει ο αποκλεισμός αυτής της ε, χώρας και να τελειώσουν οι κυρώσεις. Θεωρώ πως η πολιτική των κυρώσεων πραγματικά δεν είναι σε θέση να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Θα θέλαμε λοιπόν η διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα να οδηγήσει σε μια γενικότερη ζώνη χωρίς πυρηνικά στην Μέση Ανατολή. Επίσης θα πρέπει να ξαναξεκινήσει ο πολιτικός διάλογος σε, επίπεδα για, σε υψηλό επίπεδο για να καταλήξουμε σε μια αποκλειστικά ειρηνική και διπλωματική λύση όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. θέλω να επαναλάβω πως η κλιμάκωση και οι κυρώσεις δεν οδηγούν σε αποκλιμάκωση, αλλά στο ακριβώς αντίθετο. Η συνεχής κλιμάκωση και επέκταση των κυρώσεων είναι πολιτική κλιμάκωσης και φοβάμαι πως με την εμπειρία του Ιράκ και του τι συνέβη εκεί πέρα, θα πρέπει επιτέλους, α, ε, δεν ξέρω, ίσως να αρχίσουμε να δούμε πως αυτή η πολιτική οδηγεί σε μια στρατιωτική παρέμβαση. Θα πρέπει να δούμε και το ότι οι αποφάσεις ε, του ΟΗΕ συνέβησαν έλαβαν χώρα υπό τους περιορισμούς του άρθρου 41 που αποκλείει στρατιωτική παρέμβαση. Επίσης το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν έχει παραβιάσει τη συνθήκη μη διάδοσης ε, των πυρηνικών όπλων. Επίσης δεν έχει κυρωθεί το ε, επιπρόσθετο πρωτόκολλο από το Ιράν όπως και από άλλες χώρες. Πολλές τροπολογίες έχουν ε, τον χαρακτήρα αυτό της απομόνωσης και της κλιμάκωσης ε, της στάσης μας έναντι του Ιράν. Άρα δεν μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, κυρία Αλόζη. Ο κύριος Τάνοκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο τον κύριο Μπέλτερ, η ομάδα μου ECR συμμερίζει τη βασική του προσέγγιση έναντι αυτού του βίου Καθεστώτο, ε, Δεν μπορεί να διαβάσει όλες τις συμβαστικέ τροπολογίες του και τις τροπολογίες του γενικότερα ακόμα. Όπως και άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελα να συναντηθούν οι σκιώδεις. Εγώ είμαι σκιώδης για την ομάδα μου. Δείχνει συζήτηση της αποκλίνουσης απόψης. Όχι μόνο εντό κοινοβουλίου, αλλά και στη διεθνή κοινότητα μεταξύ εκείνων που είναι επιθετική και εκείνοι που είναι πιο φιλιρινικοί. Ο Ομπάμα έχει καλές προθέσεις. Όμως καταστροφικές οι προσπάθειές του για να τίνει χείρα βοηθείας προς αυτό το καθεστώς. Δεν κατέληξε πουθενά αυτή η προσπάθεια. Και είναι παράλογη η πρόταση της ΓΚΟΕ να μην επιβληθούν κυρώσεις και να ακολουθήσουμε μια πολιτική καθησυχασμού του καθεστώτος που έχει παραβιάσει τις συνθήκες. Έχουν μηχανήματα κεντροφυγικά για να εμπλουτίζουν το ουράνιο και αυτό είναι παραβίαση. Αν αυτό δεν επισύρει κυρώσει, ποιο ο λόγο τη συνθήκη μια διάδοση των πυρηνικών όπλων. Υποστηρίζει τη Χαμά, τη Χεσμολά, τη διεθνή τρομοκρατία. Και η Χεσμολά πρόκειται ε, να διωχθεί από τον ΟΗΕ, διότι κρύβεται πίσω από την ε, δολοφονία του Πρωθυπουργού Χαράρι ε, Χαρίρη στο Λίβανο. Οι φίλοι της Εσμπολά και εκείνοι που... Ποιος θα πιστέψει λοιπόν αυτούς που θέλουν να είναι φιλικοί προς το Ιράν. Το Ιράν απειλεί το Ισραήλ. Αντί να λέμε Ιράν, να πούμε ο πρόεδρο Αχματινετζάντ ότι απειλεί το Ισραήλ. Πώ να κάνουμε διαχωρισμό του Αχματινετζάντ όταν επικεφαλή κυβερνήσεως. πώ να το διαχωρίσει του άλλου. Δεν είναι ανώτατο πνευματικό ηγέτη αλλά δεν τον υποστήριζε ο ανώτατο πνευματικό ηγέτη, δεν τα λέει αυτά. Όταν μιλά, μιλά για το Ιρανικό καθεστώ και την κυβέρνηση. Δεν μιλά μόνο για τον εαυτό του. Δεν μιλά κανεί προσωπικά το μη κάνει επικεφαλή μια κυβέρνηση όσον αφορά τα θέματα διεθνών σχέσεων. Από τα Wikileaks ξέρουμε ότι οι πιο μετριοπαθεί χώρε στην περιοχή φοβούνται αυτό το επικίνδυνο καθεστώ. Και ίσω να ξεκινήσει ένα αγώνα δρόμου για πυρηνικό εξοπλισμό στην περιοχή τη Μεσανατολή, που θα είναι καταστροφικό για την παγκόσμια ασφάλεια. Θα πρέπει η Τουρκία ε, τελικά να πιστεί να είναι φιλικός και επικοδομητικός συνομιλητής. Είναι λυπηρό ότι στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταψήφισαν τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Αυτό είναι κατά των ε, διεθνών, της διεθνούς κοινότητας των διεθνών προδιαγραφών. Χρειάζεται εξηγήσει. Προσβλέπω στην επίσημη συνάντηση με τον εισηγητή στα πλαίσια συνομιλίων με τους Κιώδης και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε δεόντω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Σαλαφράγκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Μπέλντερ, για την προσπάθειά του και να επαναλάβω, όπως είπε και ο σκιώδης εισηγητής μας, ο κύριος Γκάλερ, την προσέγγιση μας για την έκθεση αυτή. Φυσικά δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε ε, μόνο διπλωματική φρασιολογία ε, απέναντι στο καθεστώς που εκπροσωπεί ε, το Ιράν. Θα πρέπει να κάνω μια διαυγή ανάλυση σε ό,τι αφορά το γεγονό ότι κατατέθηκαν 300 τροπολογίε. Βέβαια, οι περισσότερε κατατέθηκαν από δύο κυρίω ομάδε, του σοσιαλιστέ και του πράσινου. Που ούτω ή άλλω δεν συγκεντρώνουν πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν εξετάσουμε με προσοχή αυτές τις 300 τροπολογίες που κατατέθηκαν, διαπιστώνουμε ότι ορισμένες υιοθετούν μια πιο διπλωματική εντό εισαγωγικών προσέγγιση για μια πραγματικότητα όμως που όπως και να θέλουμε δεν μπορούμε να την ε, καλύψουμε ή να, την, ε, να της δώσουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο και σε ορισμένε περιπτώσεις ε, οι τροπολογίες αυτές δίνουν έμφαση στα πιο σε πιο σκληρέ πτυχέ ε, του Ιρανικού καθεστώτο, όπω είναι η παραβιάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίση, ε, οι τροπολογίε των φιλελευθέρων μιλούν για τη μη τήρηση τη ε, Συμφωνία Διάδοση των Πυρηνικών, για το θέμα τη θανατική ποινή, το θέμα τη δίωξη των δημοσιογράφων και ανταποκριτών, το θέμα τη δίωξη του πολιτιστικού κόσμου ή κάποιων ακαδημαϊκών και πανεπιστημιακών καθηγητών. Αν βάλουμε όλε αυτέ τι τροπολογίε, τι ομαδοποιήσουμε, περιορίζουμε σε μεγάλο βαθμό τον αριθμό του. Όπως είπε ο κύριος Γκάλερ, το ζητούμενο εδώ είναι μια συνένεση, γιατί για ένα τόσο λεπτό και ευαίσθητο θέμα όπως είναι το ζήτημα του Ιράν, που είναι από τις πιο σημαντικές μαύρες τρύπες της διεθνούς πολιτικής, θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε μια ενιαία ενωμένη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση προς τους σκιώδεις ηγητές να συνεργαστούν μεταξύ τους και να συμφωνήσουν για τη διατύπωση. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική έκκληση και συμβουλή αλλά δεν θα πρέπει να παρεκτραπούμε από τη συζήτηση από το γεγονό μόνο ότι υποβλήθησαν 300 τροπολογίε, γιατί αυτέ ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένε πολιτικέ θέσει και στάσει πολιτικών ομάδων που έχουν εύλογου λόγου, αλλά θα πρέπει να αποσπάσουν την προσοχή μα από τη σωστή εστίαση αυτή τη έκθεση και από το αξιέπαινο έργο που έχει επιτελέσει μέχρι στιγμή ο συγγετής. Σας ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα. Λίγη συζήτηση, κλείνει μάλλον τη συζήτηση ο κύριος Μάουρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω δύο παρατηρήσεις μόνο. Θέλω να ευχαριστήσω όμως τον συνάδελφο τον κύριο Μπέλτερ για τη δουλειά που έκανε. Υπάρχει πρόθεση να διεξαχθεί συνάντηση μεταξύ των σχεδόν εισηγητών και αυτές τις παρατηρήσεις τις θέτω στην διάθεση αυτής της συναντήσεως. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η γενική τοποθέτηση. Το επίκεντρο αυτή τη εκθέσεω δεν είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά η προσέγγιση Ευρωπαϊκή Ενώσεω ε, προ το Ιράν. Πιστεύω ότι ένα κομμάτι τη αξιολόγηση θα πρέπει να αφιερωθεί αν και κατά πόσα από ιστορική πλευράς Ποιο ρόλο, να δούμε ποιο ρόλο έπαιξαν κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσης αρχές του 1979 όταν επέστρεψε ο Χομείνι στο Ιράν σε σχέση ε, με το πώς θα το θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς το προσεργίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς παρουσιάζεται και η ίδια είπατε πρόσωπος έναντι του Ιράν. Υπάρχει τεράστια διαφορά με άλλα λόγια μεταξύ της σημασίας του ρόλου, του σημαντικού ρόλου που έπαιξαν κάποιε ευρωπαϊκέ χώρε κατά το παρελθόν και τη πρόθεση που υπάρχει να κρύβονται οι χώρε και να μην ε, κρίνουν τα, το τι γίνεται. Εμεί πρέπει να θέσουμε απλά πράγματα, απλά ερωτήματα όσον αφορά τα γεγονότα. Ποιο είναι το καθεστώ σήμερα. Να μην θέλουμε να απομονώσουμε ούτε τον Ιρανικό λαό και ούτε το κράτος όταν το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν κάποια ζητούμενα όμως είναι υπεύθυνο μιας απόπειρας αποσταθεροποίησεως των γειτονικών χωρών. Ιράκ. Το Ιράν είναι υπεύθυνο για την απόπειρα αποσταθεροποίησεως στο Λίβανο. Το Ιράν έχει ένα ρόλο και προσπαθεί να παίξει ηγεμονικό ρόλο έναντι χωρών του κόλπου και δημιουργεί εντάσεις με τη γειτονική Σαουδική Αραβία. Ναι ή όχι. Αυτές είναι ερωτήσεις που χρήζουν απαντήσεως. Αλλιώς αν δεν δώσουμε απαντήσεις δεν έχουμε πει τίποτα. Δεν θέλουμε να δώσουμε απάντηση και προκατηλημένη για να απομονώσουμε την κυβέρνηση του Ιράν. Αλλά ίσως για κάποια σχέδια να υποχρεώσουμε την κυβέρνηση του Ιράν να βγει από την απομόνωση στην οποία τον έφερε η ιδεολογία του και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τρόπος με τον οποίο θέτουμε ερωτήσεις απλές μπορεί να μας οδηγήσει σε απαντήσεις για περίπλοκα θέματα. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Πεγιόν. Δεν χρειάζεται μανιχιαστική προσέγγιση. Πρέπει όμως να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήσεις. Διαφορετικά θα παραγάγουμε ένα κείμενο ασήμαντο. Θα ικανοποιεί κάποιες πρεσβείες, αλλά δεν θα μπορέσει τελικά, δεν θα επιτρέψει ένα τέτοιο κείμενο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαμορφώσει την ευρωπαϊκή πολιτική. Ευχαριστώ κύριε Μάωρε. Έχουμε όμως τον κύριο Βιδαλκουάδρας και την κυρία Όμεν Ρόιτεν που θέλουν να μιλήσουν. Και με αυτή τη σειρά θα μιλήσουν. Πρώτα ο κ. Βιδαλκουάδρας και μετά η κυρία Όμεν Ρόιτεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες και ιδιαίτερα ο κύριος Σαλαφράγκα, η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Ιρανικό καθεστώς είναι από τα πιο λεπτά ζητήματα της εξωτερικής της πολιτικής. Και από κάποια άποψη εκεί παίζουμε την υπόλοιψή μας, τη φήμη μας και την, το κύρος μας και την ανάγκη επίδειξη συνέπειας ως προς τις αρχές και, την, και τις αξίες μας. Το έγγραφο του κυρίου Μπέλτερ αποτελεί ένα θαυμάσιο σημείο αφετηρίας για την προσπάθεια διαμόρφωση μια θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει να μην ξεχνάμε τις πρόσφατες εξελίξεις. Πριν από λίγες μέρες, η κυρία Νασρίν Σοτουντέκ, που είναι μία δικηγόρος, ακτιβίστρια, υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνήγορος πολιτικών κρατουμένων στο Ιράν και η μητέρα δύο ανήλικων παιδιών καταδικάστηκε σε φυλάκιση 11 ε, ετών μόνο και μόνο επειδή έκανε το έργο της η γυναίκα αυτή και μάλιστα λίγο πριν ε, το νέο έτος ο κύριος Αλίσσα Ρέμι 63 ετών εκτελέστηκε, απαχωνίστηκε μόνο και μόνο επειδή είχε κατηγορηθεί, επειδή είχε ένα γιο στο, στο, σε ένα στρατόπεδο προσφύγων στο στην Άσραφ, στο Ιράκ. Και καταδικάστηκε σε θάνατο και απαχωνίστηκε, εκτελέστηκε η θανατική ποινή. Πρόκειται για απαράδεκτες φρικαλαιότητες και μια αποτροπιστική συμπεριφορά του Ιρανικού καθεστώτος. Και μάλιστα είχαμε ε, συνυπογράψει μια δήλωση διαμαρτυρίας ε, στις 25 Νοεμβρίου 400 ευρωβουλευτές και σε αυτό το ψήφισμα για τον καταβλισμό προσφύγων του Άσραφ στο Ιράκ υπενθυμίζαμε ότι πολλοί συγγενείς ε, προσφύγων του, στον καταβλισμό αυτό είχαν καταδικαστεί από το Ιρανικό καθεστώ μόνο και μόνο επειδή επισκέφθηκαν του συγγενεί του, τα μέλη τη οικογένειά του σε αυτόν τον καταβλισμό. Και μάλιστα ο κύριο Αρέμι ήδη εκτελέστηκε, απαχωνίστηκε. Οπότε τι αυτή η διαμαρτυρία, η γραπτή διαμαρτυρία, αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τίποτα. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να αισθανθούμε οργή, αγανάκτηση, αλλά και ε, μια αίσθηση αδυναμίας και ανημποριάς, γιατί μένουμε παθητικοί μάρτυρες τέτοιων φρικαλαιοτήτων ε, χωρίς ε, να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατρανώσει τη θέση της και να ασκήσει δρυμία κριτική εις βάρος του Ιρανικού καθεστώτος. Και από ευκαιρία αυτής της έκθεσης για το Ιράν θα ήθελα να επενέσω τον κύριο Μπέλντερ για το εξαιρετικό του έργο και να απευθύνω μια έκκληση έκκληση από την Επιτροπή Εξωτερικών προς την ύπατη εκπρόσωπο, ώστε επιτέλους για μία φορά να ακούσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφανθεί και δημοσίως η ύπατη εκπρόσωπος να λάβει θέση για αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες του Ιρανικού καθεστώτος και κυρίως υπό το φω και των τελευταίων εξελίξεων, θα ήθελα η εκπρόσωπος να εκφράσει την ανησυχία της και να καταδικάσει δρυμύτατα αυτές τις επιθέσεις ε, εις βάρος των προσφύγων ε, του καταβλισμού Άσραφ εκ μέρου των ε, πρακτόρων και των εκπροσώπων του Ιρανικού καθεστώτος. Ευχαριστώ κύριε Η Κυρία Μελβάη, ήταν έχει το λόγο. Ναι κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο γιατί Μιλήσαμε μόλις για τη σχέση Ιράν-Τουρκίας και θέλω να ρωτήσω τους συναδέλφους, να καταθέσω και μία πρόταση, να δούμε την έκθεση της Τουρκίας και να δούμε τις τότε διατυπώσεις και να τις βάλουμε εδώ μέσα. Αυτό σημαίνει κύριε Πρόεδρε πως διαπιστώνουμε πως η Τουρκία παίζει έναν παραπάνω από ενεργό ρόλο στην ε, πολιτική αυτή ως ε, περιφερειακός παίκτη πρώτον. Δεύτερον, πώς θεωρούμε πως και η ύπατη εκπρόσωπος θα πρέπει να σκεφτεί καλά και σοβαρά το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή για να τον εκμεταλλευτεί και να υπάρχει κάποιος συντονισμός. Κατόπιν στο σημείο 39 λέμε πως και η Τουρκία μπορεί να βοηθήσει να προλάβουμε το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν. Μεταλυπόμαστε για το ότι η Τουρκία ψήφισε διαφορετικά στον ΟΗΕ και τέλος θα μπορούσε το τελευταίο στοιχείο να είναι να ζητήσουμε από την Τουρκία να συνεισφέρει στον εκδημοκρατισμό και την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν ε, συντονιζόμενοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν μπουν αυτά τα στοιχεία κύριε Πρόεδρε νομίζω πως ε, έτσι με έναν τρόπο ουδέτερο θα έχουμε καταφέρει να πούμε αυτό το οποίο ε, όλοι θέλουμε εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μανρόιτεν. Νομίζω ότι εδώ ο εισηγητής ο κύριος Μπέλντερ, εάν θέλει, μπορεί να μιλήσει και να σχολιάσει τις διάφορες παρεμβάσεις που ακούστηκαν πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση από αυτού του θέματος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για αυτή τη συζήτηση Νομίζω πως ε, θα μπορέσουμε να συμβαστούμε. Εντάξει, μπορεί κάποιος να έχει διαφορετικό όραμα και άποψη, αλλά δεν χρειάζεται απελπισία. Και νομίζω και με τον κύριο Πεγιόν είχαμε κάποιες διμερείς συζητήσεις. Οπωσδήποτε βεβαίω και τις μελέτες και τα διαφορά θα τα πάρω τελείως σοβαρά. Νομίζω πως ε, η Γραμματεία ήδη αυτή την εβδομάδα θα προετοιμάσει μια ημερομηνία για να μπορέσουμε να βρεθούμε όλοι μαζί. Πράγματι και η πρόταση της συγκεντρίας για την Τουρκία πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω πως ε, έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε μια καλή έκθεση και νομίζω πως ε, ο ρόλος ε, του βουλευτή είναι βεβαίως να δει που και που και το ποια είναι το πώς θα φτάσουμε στην ε, ψηφοφορία βεβαίως αλλά θα πρέπει να δούμε και με τους εισηγητές πώς θα έχουμε μια στιβαρή ομοφωνή πλειοψηφία εν πάση περιπτώσει και να πω επίσης πως και στη τελική ανάλυση είμαστε κοινοβούλιο και όχι ε, διπλωματικό σώμα. Πολύ καλά κυρία Μπέλτερ. Σε αυτή τη φάση μπορούμε να ανακοινώσουμε το χρονοδιάγραμμα για το θέμα 1η Φεβρουαρίου θα εφητηθεί στην ΑΦΕ ψηφοφορία στην Ολομέλεια προβλέπεται στην πρώτη σύνοδο του Μαρτίου του 2011. Εδώ θα πρέπει να διακόψουμε τη συνεδρίασή μας που θα συνεχίσει στις 11 με το σεμινάριο για την Ισλανδία υπό την Προεδρία του συναδέλφου του κυρίου Φιωρέλο Προβέρα. Είστε επανειδήν. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, μετά την πρωινή συνεδρίαση και τη διακοπή, συνεχίζουμε το εργαστήριο με το θέμα Ισλανδία στην Ευρωπαϊκή, Ένωση, προκλήσεις και προπτικές. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και δέχομαι θετικά το γεγονός ότι η Ισλανδία έχει παρουσία όλο και πιο συχνή ε, στην ημερήσια διατάξη της Επιτροπής αυτής και θέλουμε να υποστηρίξουμε και την υποστήριξη των υποψηφίων χωρών και των ενδεχομένων υποψηφίων χωρών. Το εργαστήριο το σημερινό εντάσσεται σε μια σειρά εκδηλώσεων που προωθεί η δική μας Επιτροπή που απευθύνεται προς αυτή τη σκανδιναβική, τη βόρεια χώρα, την Ισλανδία που είναι υποψήφια για προσχώρηση. Οι απόψει εκφράσουν σήμερα οι εμπειρογνώμονε και η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα συμβάλλουν με χρήσιμο τρόπο στη, στη διατύπωση ε, του ψηφίσματος που ε, εισηγητής ο κ. Πρέντα και θέλουμε να στείλουμε επίσημα την προσωπία μέχρι το τέλος του έτους στην Ισλανδία για να συζητήσουμε με κροσόπους του, της κυβερνήσεως, της κοινωνίας των πολιτών και του κοινοβουλίου της χώρας τα θέματα τα επίκαιρα που έχουν ε, σχέση με την ένταξη της χώρας. Για να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας όσον αφορά το θέμα και για να έχουμε ένα φόρουμ για καλό διάλογο Ετοιμάσαμε αυτό το εργαστήριο και καλέσαμε του επιφανεί καλεσμένου. Εδώ έχουμε τον κύριο Βάλντορ Τόλαλσον, καθηγητή ε, πολιτικών επιστημών ε, του Ζαν Μονέ, Πανεπιστημίου του Ρέικιαβικ, έδρα Ζαν Μονέ, που θα μιλήσει για το γενικό πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ενώσεω και Ισλανδία και ποια είναι η δημόσια συζήτηση στην Ισλανδία για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητώ συγγνώμη εάν δεν ε, προφέρω τα επίθετά σα και τα ονόματά σα σωστά. Ο Ντέιβιτ Κάρι, του τμήματος οικονομίας ε, θα εκφράσει την, το, θα αναφερθεί στα θέματα οικονομικά και χρηματοστικά ο κύριος Μπέιλς που είναι καθηγητής επισκέπτης στο Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας και το Stockholm ε, Peace Research Institute ε, θα αναφερθεί στα θέματα ασφαλείας που δημιουργούνται με την προσχώρηση της Ισλανδίας άλλες παρατηρήσεις από τον Αλεξάνδρα Γασχράντε, Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα διεύρυνσης και Νίκολα Άναγκαν ε, που είναι αντιπρόεδρος της ε, Επιτροπής για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ισλανδίας. Έχουμε και τον Γκραμ Χάνρι που είναι σύμβουλος ανώτερος του European Policy Center που μπορεί να συνοψίσει κάποια διαφορετικά θέματα για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει με τα μέλη του Κοινοβουλίου Λοιπόν, αμέσως παρευθύ δίνω το λόγο στον κύριο Μπάλντουρ Τόραλτσον που έχει το λόγο. Έχει το λόγο κύριε Τόραλτσον. Κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευκαιρία που μου δίνετε στη συμμετοχή σε αυτό το σεμινάριο. Στο Πανεπιστήμιο μου στην Ισλανδία, ένα από τα καθήκοντα που έχω είναι να εξηγήσω το θέμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στους ε, φοιτητές μου και στο κοινό. Και αυτό είναι και το αγαπημένο μου θέμα άλλωστε. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε επτά κυρίως θέματα και να καταλήξω σε σύντομα συμπεράσματα προσπαθώντας να δώσω μια απάντηση στο ερώτημα τι χρειάζεται για να είναι θετικό το δημοψήφισμα ένταξη στην Ισλανδία. Η οικονομική κρίση ξεκίνησε με την ε, καταράκωση της Ισλανδικής κορώνας το Μάρτιο 2008 και έτσι δόθηκε ένα έναυσμα για τη συζήτηση αυτή. Βέβαια, ε, αμφισβητήθηκαν και η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική της Ισλανδίας καθώς και η απροθυμία ε, της Ισλανδίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι όμως ανοίχθηκε ένα παράθυρο ευκαιρίες για τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις και το θέμα της ένταξης έγινε και το μείζον ζήτημα των εκλογών του Απριλίου του 2009. Οι σοσιαλδημοκράτες μάλιστα ε, θεώρησαν την ε, υποψηφιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως απαραίτητη, ε, απαραίτητη προϋπόθεση για την σύναψη κυβέρνηση συνασπισμού και για την δημιουργία με μια δημιουργία ενός ευρύτερου συνασπισμού και με το, ελεύθερο, ε, με το αριστερό και πράσινο κίνημα μετά τις ε, απριλινές εκλογές. Οι σοσιαλδημοκράτες πιστεύουν ότι το μέλλον της Ισλανδίας και το πεπρωμένο της Ισλανδίας βρίσκεται στο ευρωπαϊκό όραμα και την ευρωπαϊκή ολοκληρώση. Και μάλιστα ε, εντάχθηκε η Ισλανδία στην ΕΖΕΣ και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο τα υπόλοιπα κόμματα της Ισλανδίας δεν συμμερίζονται τη φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση των σοσιαλδημοκρατών. Το κίνημα αριστεράς και πρασίνων είναι αναφαδό κατά της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα πολύ απρόθυμα δέχτηκε να συμφωνήσει με την υποβολή υποψηφιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να σχηματιστεί η πρώτη κεντροαριστερή κυβέρνηση στην ε, Ισλανδία. Βέβαια υπάρχει και άλλος διχασμός στην αριστερά στην Ισλανδία. Για παράδειγμα υπάρχουν κάποιοι που είναι, ε, ήταν, τάχτηκαν υπέρ της μονομερούς εφαρμογής του ευρώ πριν της, ε, τη διεξαγωγή των εκλογών για να προσετεριστεί φιλοευρωπαίους ψηφοφόρους, ενώ άλλες ε, αριστερές παρατάξεις είναι υπέρ της απόσυρσης από ψηφιότητες για την ε, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν λοιπόν διστάμενες απόψεις όπως βλέπετε. Πριν από δύο χρόνια ε, το μεγαλύτερο κόμμα την πολιτική του, είναι επίσημα υπέρ της υποψηφιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με προϋποθέσεις όμως και μάλιστα δύο τρίτα των ε, βουλευτών αυτού του κόμματος καταψήφισε την υποψηφιότητα. Επίσης ε, και οι βουλευτές του κινήματος ε, των πολιτών που συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες του προηγούμενου χειμώνα είναι αρκετά σκεπτικιστές ως προς την προοπτική ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτικές συζητήσεις στην Ισλανδία κυριαρχήθηκαν ε, από τις ε, συζητήσεις για το iSave. Επίσης ε, αναλύθηκαν τα πλεονεκτήματα μιας υποψηφιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες να προωθήσουν τη θέση τους γιατί υπάρχει ένας αναρχόμενος εθνικισμός στην Ισλανδία και η, η Ισλανδία θεωρούν ότι εκτός αν εξαιρέσουμε τις συνήθειες Φερόες, οι υπόλοιποι τους έχουν εγκαταλείψει γειτονικές χώρες στη στιγμή της μεγαλύτερης ανάγκης τους. Η κατάσταση κοινή γνώμη ότι αφορά την υποψηφιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάστηκε από το θέμα της συζήτησης για το Ice Save. Και μάλιστα από τον Απρίλιο 2009 οι περισσότεροι ψηφοφόροι τάχθηκαν κατά της ένταξης. Ε, έτσι φάνηκε από τι δημοσκοπήσεις. Σε αντίθεση με την προηγούμενη δωδεκαετία, όπου σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν μια πλειοψηφία των Ισλαδών υπέρ τη ένταξη. Και μάλιστα το καλύτερο αποτέλεσμα φάνηκε μετά την οικονομική κατάρρευση. Βέβαια, οι περισσότεροι πολίτες είναι υπέρ τη συνέχιση των ενταξιακών συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το περασμένο έτος φάνηκε μια τάση για απόσυρση της υποψηφιότητας, αλλά αυτή η τάση φαίνεται ότι έχει ξοβελιστεί. Η συζήτηση πάντως για την ένταξη αρχίζει και αποκτά μια καλύτερη ισορροπία και μπαίνει σε μια οδό εμβάθυνσης. Μάλιστα υπήρξε μια, ένα κίνημα για το όχι, κυρίως στην Ήπεθρο και ιδιαίτερες κοινότητες γεωργών και αλλιέων. Αυτή ήταν η περισσότερη ε, πιο έντονη πολέμη της ένταξης της Ισλανδίας. Μάλιστα και στο Κοινοβούλιο έχουν υποβληθεί ψηφίσματα για τη διοργάνωση δημοψηφίσματος ό,τι αφορά τη συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ή μερικές φορές ζητήθηκε και η άμεση απόσυρση της Ισλανδικής αποψηφιότητας ε, για ένταξη. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν ε, ε, διαμορφώθηκε θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς τις προτάσεις αυτές. Βέβαια το κίνημα του όχι στηρίχθηκε και στην ε, ε, αντίδρασή του ως προς την συμπερίληψη του κοινοτικού κεκτημένου και πριν την ένταξη της Ισλανδίας. Μάλιστα η Ισλανδική κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι πριν ληφθεί οριστική απόφαση για την υποψηφιότητα δεν πρόκειται να γίνει προσαρμογή με το κοινοτικό κεκτημένο και σε καμία περίπτωση πριν την διεξαγωγή σχετικού δημοψηφίσματος. Τώρα το φιλοευρωπαϊκό κίνημα ανασυντάχθηκε και μάλιστα ε, ίδρυσε και μία οργάνωση με τον τίτλο «Ισχυρότερη Ισλανδία, ένα έθνος μεταξύ άλλων εθνών». Και μάλιστα έχει ιδιαίτερη υποστήριξη γύρω από την πρωτεύουσα, το Reykjavik, και έχει δεχτεί την υποστήριξη πολλών συνδικάτων και των κομμάτων των συντηρητικών, των σοσιαλδημοκρατών και των προοδευτικών. Ο επιχειρηματικός κλάδος και πολλά συνδικάτα έχουν μέχρι στιγμής σιωπήσει για το θέμα το ευρωπαϊκό μετά την αρχική τους ε, υποστήριξη της ε, Ισλανδικής υποψηφιότητας. Φαίνεται όμως ότι θα επανέλθουν στη συζήτηση όσο πλησιάζει η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για την υποψηφιότητα. Πάντως, η Συνομοσπονδία των Ισλανδών Εργοδοτών δεν συμμετέχει ενεργά στην συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιτία ε, της διχόνοιας που υπάρχει στο Διοικητικό της Συμβούλιο, γιατί ε, οι Ισλανδοί εφοπλιστές ε, που είναι και η κρατούσα δύναμη στην Ομοσπονδία των Εργοδοτών, είναι κατά τις υποψηφιότητες και μπορεί να δημιουργήσει ένα, μια αναχέτηση και μια ανασχετική ψήφο σε ό,τι αφορά την ε, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γίνονται πολλές συζητήσεις σε ό,τι αφορά τα υπέρ και τα κατά της ε, ένταξης της Ισλανδίας, αλλά δυστυχώς ε, δεν συμμετέχουν αρκετοί εμπειρογνώμονε στι συζητήσει αυτές. Και μάλιστα μια σημαντική εφημερίδα είναι υπέρ τη υποψηφιότητα και στα βασικά της άρθρα τάσεται υπέρ τη ένταξη, ενώ μια άλλη πιο συντηρητική εφημερίδα οργανώνει μια δρυμία εκστρατεία ει βάρο της υποψηφιότητα, κατά της υποψηφιότητα, με επιχειρήματα κυρίω την αλία. Πάντως τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πιο ισορροπημένα στη θέση τους, αλλά θα μπορούσαν να ταχθούν πιο δραστήρια υπέρ της ενημέρωσης του κοινού για το θέμα της υποψηφιότητας. Τώρα, ποια θα είναι η έκβαση του δημοψηφίσματος, θα είναι θετική. Για, μια, για την υιοθέτηση μιας ενταξιακή συνθήκης και για να εγκριθεί από την πλειοψηφία των ψηφοφόρων θα πρέπει να διασκεδαστούν οι ανησυχίες τους ό,τι αφορά δύο βασικά στοιχεία καταρχήν την ικανοποιητική συνέχιση των ελευτικών δραστηριοτήτων της Ισλανδίας και της διαχείρισης των χωρικών της υδάτων και στα πλαίσια της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Και δεύτερον, το θέμα της προστασίας της αγροτικής κοινότητας της Ισλανδίας στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι δύο ανησυχίες θα πρέπει να διασκεδαστούν. Ένα άλλο θετικό ζήτημα σε μια συμφωνία θα ήταν μια σταθεροποίηση μια συμφωνία σταθεροποίηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα τη Ισλανδική κορώνα και να ε, πληρωθούν από την Ισλανδία τα κριτήρια για την ε, εισαγωγή του ευρώ. Αν εκπληρωθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, πιστεύω ότι η κυβέρνηση, τουλάχιστον οι σοσιαλδημοκράτες, θα μπορούσαν να έχουν πιο ε, πιστικά επιχειρήματα και να κερδίσουν το δημοψήφισμα για μια θετική έκβαση του Ισλανδικού Δημοψηφίσματος για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα αν φανεί το στρατηγικό συμφέρον της Ισλανδίας για την πλήρη ένταξή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, τι θα γίνει με τα άλλα κόμματα, θα συνεχίσουν την αντίστασή τους. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προβλέψουμε την ε, μελλοντική του θέση. Πάντω ε, εμεί στην Ισλανδία ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μας βοηθήσουν με την κατανόηση και την υποστήριξή τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Τόλβαρσον. Πάρα πολύ σαφής η παρουσίασή σας. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Άλισον Μπέιλς. Μάλλον δεσποινής Άλισον Μπέιλς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε καθώς προβάλλεται η παρουσίασή μου να πω πως είναι πάντα τιμή να με προσκαλείτε να μιλήσω εδώ στο Κοινοβούλιο και όπως και ο φίλος μου ο κύριος Μπάλτερ θα σας δώσω και εγώ βασικές πληροφορίες γιατί η Ισλανδία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα και είναι ενδιαφέρον να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Ε, ίσως το πιο προφανές είναι πως ήταν βεβαίως ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχει ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχουν πρακτικοί λόγοι γι' αυτό. Σε ένα τόσο απομένομενο νησί οι χερσαίες επιχειρήσεις είναι απίθανες και η ασφάλεια της Ισλανδίας ουσιαστικά βασίζεται σε αεροναυτική κάλυψη και είναι δύσκολο για ένα έθνος 300.000 ανθρώπων να έχει κάτι τέτοιο όμως το να μην έχει ενοπλές δυνάμεις είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό στην πολιτική κουλτούρα της Ισλανδίας. Ταιριάζει με το ότι είναι ένα σχετικά νέο κράτος. Έλεγξε πλήρως την εξωτερική της πολιτική το 1944 και ήθελε βεβαίως να αποτελέσει μια ειρηνική δύναμη. Μάλιστα νομίζω πως η Ισλανδία θα προτιμούσε την ε, ουδετερότητα, αλλά στον ψυχρό πόλεμο βεβαίω βρέθηκε σε μια εκτεθειμένη στρατηγική θέση στο Βόρειο Ατλαντικό. Η μόνη λύση, η πρακτική ήταν να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ο μόνος τρόπος για να την υπερασπιστεί το ΝΑΤΟ ήταν μέσω των δυνάμεων των ΙΠΑ από την Δύση που κατέλαβαν μια μεγάλη βάση στο Κέπλαβικ και βεβαίως ε, παρήχαν και άμυνα και πολλέ χρήσιμε υπηρεσίε για την Ισλανδία. Το ΝΑΤΟ προσωπούταν από ένα μεγάλο ραντάρ αεράμυνα, επίσης στο Κέπλαβικ, αλλά όσο ήταν εκεί η ήπα φρόντιζαν και αυτά τα ραντάρ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις, όπως ξέρετε, αποσύρθηκαν μονομερός ε, το 2006 και θα επανέλθουμε αργότερα στα αποτελέσματα που είχε αυτή η κίνηση. Προς στιγμήν όμως καλό είναι να σκεφτούμε το τι σημαίνουν αυτές οι εμπειρίες για το πώς αντιλαμβάνεται την άμυνα και την ασφάλεια η χώρα. Η άμυνα ουσιαστικά ήταν κάτι που έκαναν κάποιοι άλλοι. Αυτό ήταν πάντα κάτι το επίμαχο και υπήρχαν βεβαίως αντιδράσεις στην παρουσία, είπα, και το ειδικά από την ε, ριζοσπαστική αριστερά. Ως αποτέλεσμα αυτού, ε, αυτά τα οποία έκανε η ίδια η Ισλανδία, δηλαδή αποτελεσματική ακτοφυλακή, έρευνα και διάσωση και ε, συνήθη της πολιτικής άμυνας δεν ορίζονταν υπό τον όρο άμυνα και ασφάλεια. Δίνονταν έμφαση στον πολιτικό του, στον μη στρατιωτικό χαρακτήρα. Και η Ισλανδία δεν χρειαζόταν να αναπτύξει μία έννοια ε, ασφάλειας ε, γιατί βεβαίως δεν είχε μεγάλη συγκρούση σε έγκλημα 80% αυτάρκεια στην ενέργεια και βεβαίως ε, είναι πιθανότερο να κερδίσει στις πρώτες φάσεις της κλιματικής αλλαγής. Αλλά μετά την απόσυρση των ήπα έπρεπε οι ηγέτες της Ισλανδίας να σκεφτούν τι θα κάνουν για την ασφάλειά τους. Να διατηρήσουμε βεβαίως κάποια για να διατηρήσουν κάποια αμυντική προστασία έκαναν διμερεί συμφωνίες με Νορβηγία, Δανία και κάποιες άλλες χώρες και το ΝΑΤΟ συμφώνησε να αναπτύσσει ad hoc στρατεύματα από καιρού καιρών για να επιδεικνύει την ε, δυνατότητά του να βοηθάει στην αέρα της Ισλανδίας. Επίσης υπάρχει ένα νέο σκάφος της ακτοφυλακής και βεβαίως ε, υπήρχε η σκέψη στο Κέπλαβικ να υπάρξει Ισλανδική υπηρεσία άμυνας, κάτι όμως το οποίο ήταν επίμαχο για αριστερά και δεξιά και η υπηρεσία δεν θα συσταθεί και το έργο θα το αναλάβουν άλλες υπηρεσίες. Ακόμα αυτά συζητώνται Από ό,τι φαίνεται, το περισσότερο έργο θα πάει στο Υπουργείο των Εσωτερικών και πιθανώς το Φυλακή. Γενικά, όσον αφορά τον ορισμό της ασφάλειας, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία υπό την προηγούμενη κυβέρνηση που ήταν δεξιά, συνασπισμός δεξιάς και σοσιαλδημοκρατών, ήταν να ζητηθεί μια ανεξάρτητη ανάλυση κινδύνου και η έκθεση αυτή που δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 2009 για πρώτη φορά παρουσίασε μια ευρύτατη προσέγγιση της ασφάλειας και προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν από πλευράς Ισλανδίας, π.χ. οικονομική ασφάλεια, ηλεκτρονική ασφάλεια, περιβαλλοντική ασφάλεια κτλ. Δεν ανελήφθη κάποια άμεση δράση, αλλά η τωρινή κυβέρνηση υποσχέθηκε στα μέσα του 2010 να αναπτύξει μια στρατηγική εθνικής ασφάλειας που θα βασίζεται μάλλον σε αυτή την αξιολόγηση κινδύνων. Όσον αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διαπραγματεύσεις, νομίζω πως όσα βλέπετε στη διαφάνεια είναι απλά πράγματα, δεν αναμένουμε σοβαρά προβλήματα. Για να μπει πλήρως στην ΚΕΠΑ και στην ΕΠΑΑ η Ισλανδία. Ε, η Ισλανδία έχει ευρωπαϊκά ιδεώδη, θα έλεγα σκανδιναβικές αξίες ε, της παγκόσμιας αροχής, ε, αφοπλισμού και υποστήριξης ειρηνευτικών αποστολών. Έχει συμμετάσχει σε ειρηνευτικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολιτικές δυνάμεις, ειδικού δηλαδή που αποστολές που οργανώνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Οπωσδήποτε η Ισλανδία θέλει να ξεκαθαρίσει πως μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω ένα μη στρατιωτικό κράτο και δεν σκοπεύει να αποκτήσει ενόπλες δυνάμεις στο μέλλον. Τώρα, ο στρατηγικός ρόλος της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς ε, τον βλέπουν στην Ισλανδία. Ακριβώς επειδή η βασική έννοια της ασφάλειας και της άμυνας είναι κάτι τόσο στενό, ακριβώς μια μειοψηφία συνειδητοποιεί μέχρι στιγμής πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, είναι στρατηγική δύναμη, μπορεί να προστατεύσει στρατηγικά την Ισλανδία και κυρίως να την προστατεύσει οικονομικά και να επιβάλλει και μια οικονομική πειθαρχία. Και αυτούς οι οποίοι πιέζουν για να ενταχθεί η Ισλανδία, αυτή η στρατηγική κάλυψη από την Ένωση, επιπροσθέτως βεβαίως προς την κάλυψη του ΝΑΤΟ, νομίζω είναι ένα ισχυρό επιχείρημα. Από πλευράς τώρα της Ένωσης, η Ισλανδία δεν είναι καμία, ένας μεγάλος στρατηγικός πόρος, ούτε και στρατηγικό βάρος. Τα στρατηγικά ζητήματα οπωσδήποτε δεν συγκρίνονται με τη διεύρυνση των Δυτικών Βαλκανίων. Αλλά υπάρχει ένα ενδιαφέρον ζήτημα και αυτό βέβαια αφορά το άνοιγμα της Αρκτικής γιατί όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει την πολιτική της στην Αρκτική και σκοπεύει να παίξει ένα ρόλο εκεί ειδικά στο πλαίσιο κλιματικής αλλαγής και οικονομίας και στο πλαίσιο αυτό η θέση της Ισλανδίας και η και το γεγονό ότι είναι κοντά στην Αρκτική ε, είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γενικά νομίζω είναι σε καλή θέση η Ισλανδία για να αποτελέσει θετικό εταίρο. Έχει εξαιρετικές σχέσεις με τους γειτονέ της, ε, έχει σκανδιναβική συνεργασία και νιώθει ιδιαίτερα κοντά στην Γαριλανδία και τις Φαρόες νήσους και έχει ένα ε, ιδιαίτερο δίκτυο συνεργασίας μαζί τους. Ταυτόχρονα έχει πολύ χαλαρές σχέσεις με τη Ρωσία, κάτι το οποίο δεν διαταράχτηκε από κάποιες ανησυχίες ε, περί ρωσικών αεροσκαφών που πλησιάζουν περισσότερο την Ισλανδία. Οι γενικές σχέσεις είναι θετικές και τέλος η αρκτική πολιτική της Ισλανδίας είναι λίγο πολύ ε, στις γραμμές της πολιτικής της Ένωσης και τονίζω εδώ πέρα πως η Ισλανδία στηρίζει την Ένωση ε, στο να έχει έναν ισχυρότερο ρόλο στο Αρκτικό Συμβούλιο. Ήδη συνεργάζονται οι δύο πλευρές ε, ως προς αυτό και θα συνεχίσουν να συνεργάζονται και χωρίς την ένταξη, αλλά και θα ήθελα να τελειώσω εδώ πέρα κυρίως λόγω του αρκτικού παράγοντα, ακόμα και αν η άμυνα της Ισλανδίας δεν στενίζεται άμεσα, δεν σχετίστηκε άμεσα στο παρελθόν με την ε, διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο με δυναμικό τρόπο από το πώς αλλάζει η ασφάλεια στη δική μας περιοχή του κόσμου και τα νέα πεδία αναμέτρησης που ανοίγονται. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο David Κάρι τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω για κάποιες οικονομικές σηματοδοτικές πτυχές που αφορούν το αίτημα της Ευρωπαϊκής Ενώσης να, της Ισλανδίας να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να εστιαστώ επί τριών θεμάτων Πρώτα φορά προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπει η χώρα στην Ευρωζώνη. Δεύτερον, δύο βασικά θέματα στις διαπραγματεύσεις που αφορούν την κοινή αλληλευτική πολιτική και την κοινή αγροτική πολιτική. Και τρίτον, συμμόρφωση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης Γιατί ζήτησε ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ισλανδία ήθελε να μπει στην Ευρωζώνη ουσιαστικά. Η οικονομική κρίση έγινε πιο σοβαρή λόγω της έλλειψης προσβάσεως στην δανειοδότηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Σχετικής Τράπεζας. Όμως οι τράπεζες της Ισλανδίας είχαν περιορισμένη πρόσβαση στα διάφορα μέσα ενίσχυσης μέσω των θηγατρικών τους στην Ευρωζώνη. Αλλά πιο σημαντικό, είχαν προβλήματα ρευστότητας οι της Ισλανδίας διότι θεωρούνται αφαιρέγγιες και αυτό τις εμπόδισε από τις αγορές δαδιοδότησης μεγάλων ποσών. Και αυτό επιβεβαιώθηκε και από την κλίμακα των απολειών όταν χρεοκόπησαν τράπεζες τον Οκτώβριο του 2008. Όμως, παρά τα αυτά, μια θετική πτυχή το ότι είχαν δικό τους νόμισμα ήταν ότι η υποτίμηση του νομίσματος διευκόλυνε προσαρμογή της πραγματικής οικονομίας μετά την οικονομική κρίση. Βλέπουμε στο γράφημα ότι οι εισαγωγέ αμερίδιο μερίδιο της γενικής ζήτησης μειώθηκαν σημαντικά και εξαγωγέ σαν μερίδιο του ΑΕΠ αυξήθηκαν σε ποσοστό του ΑΕΠ. Επόμενο γράφημα, απώλειες ανταγωνιστικότητας. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής άνθησης ε, αντεστράφησαν όλα τα πλεονεκτήματα από αυτή την κρίση και την υποτίμηση. αν ήταν στην Ευρωζώνη δεν θα έκανε τη μεγάλη διαφορά στην κλίμακα της οικονομικής κρίσης που πέρασε η Ισλανδία. Όμως, έχει πολλά ωφέλη για την Ευρωζώνη, ε, για την Ισλανδία Ευρωζώνη. Θα αυξηθεί το εμπόριο με τις χώρες Ευρωζώνης, αν μπει στην Ευρωζώνη. Θα μειωθούν τα επιτόκια στην Ισλανδία θα μειωθούν οι, τα ασφάλιστρα για τους ε, ε, κινδύνους του νομίσματος. Οπότε θα υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως, αν μπει στην Ευρωζώνη η Ισλανδία. Δεν είναι στην καλύτερη δυνατή περιοχή στον αφορά το νόμισμα. Κοιτάξτε τον πίνακα. Συντελεστή συσχετισμού δείχνουν διαταραχές μεταξύ Ευρωζώνης και Ισλανδίας. Η ζήτηση έχει μικρό σχετισμό και οι κλονισμοί όσον αφορά την παροχή, την προμήθεια δεν επηρεάζεται καθόλου. Στον ζώντιο άξονα βλέπουμε τις μεταβολές όσον αφορά την προσφορά και στον κάθετο όσον αφορά τη ζήτηση. Στο πρώτο τετραγωνίδιο, στο πρώτο πλαίσιο βλέπετε ότι η Ισλανδία δεν έχει σχετισμό για διαταραχές όσον αφορά την παροχή εμπορευμάτων προς την Ευρωζώνη και όσον αφορά τη ζήτηση είναι μικρότερες οι διακυμάνσεις. Καλύτερα θα ταιριάζαμε τη Σουηδική κορώνα η Ισλανδία. Και στο δεξιό πλαίσιο βλέπουμε ότι η Ισλανδία δεν είναι τόσο καλά προσαρμοσμένη για να είναι στην Ευρωζώνη όσον αφορά το νόμισμά της. Εν συγκρίση με άλλες χώρες όπως είναι η Γαλλία και η Γερμανία. Όμως, μια χώρα σαν την Ισλανδία μπορεί να τα καταφέρει στην Ευρωζώνη, διότι έχει πολύ ευέλικτε αγορές εργασία. Έτσι, μπορεί να κάνει τέτοιε προσαρμογές πραγματικής οτιμία που πρέπει να κάνει. Χωρίς να χαθούν θέσει απασχόλησης και παραγωγικότητα. Το μεγάλο θέμα τώρα, το δύσκολο προς διαπραγμάτευση, είναι η αλία. Η Ισλανδία έχει καλό ιστορικό στον τομέα αυτό όσον αφορά τη διαχείριση των λευτικών πόρων, βιώσιμη διαχείριση. Αν δείτε εδώ το πρώτο πλαίσιο, βλέπετε ότι τα λιεύματα στην Ισλανδία ακολουθούν στενά τις επιστημονικές προτάσεις για την αλληλεία, τη βιώσιμη του Βακαλάου. Ενώ για τη Βόρεια Θάλασσα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Εκμετάλλευση των Θαλασσών πρότεινε μορατόριο όσον αφορά αυτόν τον πόρο από το 2001 και συνολικό αλίευμα που επιτρέπεται είναι πολύ μεγαλύτερο από το μηδέν και τα πραγματικά αλιεύματα ήταν ακόμα πιο πολλά. Στην Ισλανδία όλα τα αλιεύματα πρέπει να εκφορτώνονται. Αυτό δεν ισχύει όμως στην αλία του Βακαλάου στη Βορεια Θάλασσα. Γιατί γίνεται σωστή διαχείριση αλίειας και δεν γίνεται υπεραλίευση στην Ισλανδία είναι το μεταφερό, η μεταφερόμενη ποσόστοση. Υπάρχουν δικαιώματα διοκτησία στον λευτικό τομέα και δεν θέλουν οι πόροι τους να υπεραλίευονται. Για να παραμείνει... Α, να πούμε κάτι άλλο. Η είναι πολύ σημαντική για την Ισλανδία. 40% του, του εμπορεύματος που εξάγεται, 8 και 9% του ΑΕΠ, αντιπροσωπεύει. Θα είναι σημαντικό λοιπόν για την Ισλανδία να τηρήσει την αξία του πόρου αυτού του αληφτικού. Και τα συνολικά επιτρεπτά αλλιεύματα θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικέ συστάσει. Η ιδιοκτησία, τα δικαιώματα, τα ιδιωτικά πρέπει να διατηρηθούν ε, και θα πρέπει οι ποσοστώσει να εφαρμόζονται με κάθε αυστηρότητα. Άλλο σημαντικό θέμα στι διαπραγματεύσει. Η κοινή γεωργική πολιτική, η κοινή αγροτική πολιτική και ένταξη στην ΚΑΠ. Βλέπετε τα γραφήματα. Η προστασία της γεωργίας είναι πολύ ψηλή στην Ισλανδία. Από οικονομική έποψη λοιπόν, η ένταξη στην ΚΑΠ θα είναι αποτελεσματική για την Ισλανδία. Θα μειωθεί η προστασία η αγροτική στα επίπεδα της Ευρωπαϊκή Ενώσεως και θα μεταφερθούν πόροι σε πιο παραγωγική χρήση. Θα μειωθούν οι τιμές των τροφίμων που αυξάνονται κατά 50% λόγω των πολιτικών γεωργικής προστασίας και θα μειωθούν ε, θα μειωθεί μεταφορά κονδυλίων του προπολογισμού στους γεωργούς. Δεν είναι πρόβλημα πολιτικό στην Ισλανδία. Οι πολιτικοί προσπαθούν να διαπραγματευτούν συμφωνία για να παραμείνουν υψηλά τα επίπεδα της προστασίας για τους γεωργούς. Άλλο θέμα που προανέφερα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν είναι η Ισλανδία, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα σύμφωνα σταθερότητα και ανάπτυξη. Αυτό δεν πρέπει να είναι πολύ δύσκολο για τη χώρα. Είχε καλή φορολογική πολιτική και οικονομική πολιτική πριν την κρίση και εφαρμόζει αυστηρότατο πρόγραμμα εξυγίανσης στα πλαίσια των διευθετήσεων με το Διεθνές Μεσματικό Ταμείο. Άρα θα έχουν πλεόνασμα φέτος και γενικό πλεόνασμα θα επιτευχθεί μέχρι το 2013 και το χρέος σαν ποσοστό του ΑΕΠ μειώνεται σε φωτοσχέδιο από φέτο. Θα πρέπει να είναι 15% του, κατά 15% του ΑΕΠ χαμηλότερο μέχρι το 2014. Για το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη θετικό, μπορεί να διατηρηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία στο μέλλον από τη στιγμή που θα λήξει το πρόγραμμα του Δουνουτού. ποιο είναι το συμπέρασμα, ότι η προσχώρηση είναι ελκυστική για την Ισλανδία. Αν προστατευτούν οι ελευτικοί πόροι. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο τώρα. Αλεχάνδρα Κασχράνθε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία μου στο σημερινό σεμινάριο και θα σας κάνω κάποια γενικά σχόλια σε σχέση με αυτά που ακούσαμε, χωρίς να επικεντρωθώ όμως σε συγκεκριμένη παρουσίαση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή που δίνετε στο θέμα αυτό και για τη διοργάνωση αυτού του σεμιναρίου. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή τη συζήτηση για την Ισλανδία σήμερα. Θα ήθελα να σας πω καταρχήν για ποιο λόγο θα πρέπει να δώσουμε έμφαση αυτή την έλξη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισλανδίας. Ο λόγος αυτός βρίσκεται στα άρθρα 49 και 32 της ε, συνθήκης που το πρώτο προβλέπει ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκό κράτος ε, τηρεί τις αξίες ε, του άρθρου 2 και έχει τη δέσμευση να τις προωθήσει μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το άρθρο 2 προβλέπει ότι η Ένωση στηρίζεται στις αρχές και αξίες σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κράτους δικαίου, ισότητας, αξιοπρέπειας, ε, σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Όλες αυτές οι αξίες είναι κοινέ στα κράτη-μέλη που έχουν κοινωνίες δίκαιες, με αλληλεγγύη, πλουραλιστικές και που χαρακτηρίζονται από ισότητα μεταξύ ανδρών και, ανδρών και γυναικών. Η Ισλανδία, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πληρεί πλήρως αυτές τις προϋποθέσεις ένταξης. Νομίζω ότι συμφωνούμε ως προς αυτό και είναι ένας θαυμάσιος και εύλογο λόγο που δείχνει την αμοιβαία έλξη Ισλανδία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ευρωπαϊκά μάλιστα θεσμικά όργανα αναγνώρισαν αυτό το λόγο όταν συνέταξαν την έκθεση για την ε, υποβολή υποψηφιότητα για ένταξη τη Ισλανδίας και εξετάζοντα το θέμα και υπό το πρίσμα των κριτηρίων τη Κοπεχάγης καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ήδη η Ισλανδία πληρεί τα πολιτικά κριτήρια και ήδη πληρεί και τα οικονομικά κριτήρια. Μάλιστα, η Ισλανδία πλήρει και ένα μεγάλο τμήμα και του κοινοτικού κεκτημένου. Γιατί από το 1995 και μετά ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και ως τέτοιο μέλος ήδη εφαρμόζει ένα μεγάλο τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ποσοστό, πάντως σίγουρα ένα μεγάλο τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου. Σίγουρα θα πρέπει να εφαρμόσουμε τη διαδικασία διεξοδικού ελέγχου και screening πριν την ένταξη για να δούμε αν υπάρχουν ατέλειες ό,τι αφορά την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου. Πάντως σας διαβεβαιώ ότι ήδη η Ισλανδία εφαρμόζει ένα μεγάλο τμήμα του. Τώρα εξετάζοντας όλα αυτά υπό τη σκοπιά των προκλήσεων και των προοπτικών ένταξης τη Ισλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να σα εξηγήσω ποιε κατά τη γνώμη μου είναι οι βασικέ προκλήσει. Οι βασικέ προκλήσει αφορούν κυρίω το κοινοτικό κεκτημένο, η γνωμοδότηση, η έκθεση πρόοδου και το συνεχόμενο screening για τα 33 κεφάλαια ένταξης δείχνουν ήδη αυτό που είχαμε υποψιαστεί. Ότι δηλαδή η Ισλανδία πληρεί ένα μεγάλο τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου και έχει ελάχιστα προβλήματα σε λίγα μόνο κεφάλαια. Και ποια είναι τα επίμαχα κεφάλαια? Είναι το γεωργικό κεφάλαιο, το κεφάλαιο της ελίας, το θέμα του περιβάλλοντος. Αυτά είναι τα τρία βασικά κεφάλαια στα οποία η Ισλανδία αντιμετωπίζει προβλήματα. Βέβαια εδώ ακούσαμε και για το θέμα της ασφάλειας και της ε, ένταξης στην ΚΕΠΑ. Αυτό δεν είναι προβληματικό κεφάλαιο. Είναι θέμα ετοιμότητας απλώς και προετοιμασία για την ένταξη. Η αελία όμως θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το πιο ευαίσθητο θέμα των διαπραγματεύσεων με την Ισλανδία. Ακούσαμε ήδη ότι η Ισλανδία εφαρμόζει μια προηγμένη στρατηγική διαχείριση ΑΕΛΙΑ και ενδιαφέρεται φυσικά για μια πολιτική αηφόρου διαχείριση ε, στα θέματα αλίας, αλλά θα πρέπει η Ισλανδία να ανοίξει τον αλληλευτικό της κλάδο και να τηρήσει το κοινοτικό κεκτημένο σε ό,τι αφορά το δικαίωμα εγκατάστασης, ε, την ελεύθερη ε, κυκλοφορία κεφαλαίων και υπηρεσιών, κάτι που δεν ισχύει στην Ισλανδία για τον αλληλευτικό κλάδο και κάτι τέτοιο προποθέτει ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις στην Ισλανδία. Πάντως για την κοινή αλληλευτική πολιτική ε, γνωρίζετε τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν η Ισλανδία θέλει να ενταχθεί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εστερνιστεί το νέο κοινοτικό αλληλευτικό κεκτημένο. Αλλά και η Γεωργία είναι κάπως προβληματικό κεφάλαιο, αλλά κάπως διαφορετικό από την Αλία. Θα πρέπει και εκεί να προετοιμαστεί η Ισλανδία για να ευθυγραμμιστεί με την κοινή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να θεσπίσει τα απαραίτητα όργανα, θεσμικά όργανα που προποθέτει μια τέτοια κοινή γεωργική πολιτική. Ακούσαμε ότι η Ισλανδία δεν θέλει να ευθυγραμμιστεί με το κοινοτικό κεκτημένο πριν την ένταξη. Και αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα ετοιμότητά τη ω προ την ένταξη. Γιατί αν κανεί δεν θέλει να προετοιμαστεί ε, για την ένταξη πριν να διοργανώσει το δημοψήφισμα, θα μείνει πίσω. Αλλά είναι διαφορετική αυτή η πρόκληση. Δεν είναι τόσο πρακτική πρόκληση, αλλά πολιτική. Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, η εμπορική φαλαινοθυρία που εφαρμόζεται στην Ισλανδία είναι ασύμβατη με το κοινωτικό κεκτημένο. Και επίσης υπάρχει και το θέμα της ε, επανάληψης της φαλαινοθυρίας στα πλαίσια της ε, παγκόσμιας ε, οργάνωσης για το θέμα αυτό. Αλλά αυτά τα θέματα θα συζητηθούν ε, επισταμένως. Πάντως αυτές οι βασικές προκλήσεις κοινοτικού κεκτημένου μπορούν να υπερκεραστούν. Κατά τη γνώμη μας, ναι, μπορούμε να ε, υπερκεράσουμε αυτές τις προκλήσεις. Αυτό που απαιτείται είναι η πολιτική βούληση της Ισλανδικής κυβέρνησης και σε τελικό βαθμό φυσικά και της Ισλανδικής κοινωνίας να υποστηρίξει την κυβέρνηση και τις επιλογές της. Θα ήθελα τώρα να πω δύο λόγια για τις άλλες προκλήσεις που δεν αφορούν άμεσα το κοινοτικό κεκτημένο. Η βασική είναι η οικονομική κατάσταση στην Ισλανδία και το δεύτερο είναι το ISAVE, η διάσωση του πάγου. Για την οικονομική κατάσταση αναφέρθηκε ότι το πρόγραμμα ανάκαμψης έχει ήδη εφαρμοστεί και μάλιστα έχει εγκριθεί, Μάλλον αυτή τη βδομάδα εγκρίνεται και η, η δεύτερη δόση για τη διάσωση της Ισλανδίας υπάρχει μια εμφανής βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και μάλιστα υπάρχει και το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ισλανδίας, Ολλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου και ελπίζω να εγκριθεί η συμφωνία αυτή από το Ισλανδικό Κοινοβούλιο και να εφαρμοστεί. Αυτές οι δύο προκλήσεις πάντως είναι προσωρινές, εφήμερες και πιστεύω ότι θα διεκπαιρεωθούν αυτά τα θέματα ε, πολύ σύντομα. Και το θέμα βέβαια του σκόβρου είναι ένα πρόβλημα στην Αλία που θα πρέπει να διαθετηθεί το συντομότερο δυνατό. Πάντως πιστεύω ότι η Ισλανδία θα πρέπει να βελτιώσει την επικοινωνία της και με τους πολίτες και να τους ενημερώνει πιο εμπεριστατωμένα για το θέμα της διεύρυνσης. Αλλά αυτό είναι ευθύνη της Ισλανδικής κυβέρνησης. Θα πρέπει να αναβαθμιστεί η συζήτηση για την ένταξη στην Ισλανδία. Θα ήθελα τώρα να πω δύο λόγια και για τις προοπτικές της Ισλανδικής ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση αυτά που είπαμε μπορούμε να καταλήξουμε εύκολα στο συμπέρασμα ότι οι προοπτικές της ένταξης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θαυμάσιες. Κατά πάσα πιθανότητα είναι πολύ καλύτερες οι προοπτικές για την Ισλανδία από ό,τι για οποιοδήποτε άλλη χώρα που προσβλέπει στην προσχώρηση. Βέβαια, τι θα συμβεί στην πράξη, μόνο η Ισλανδία μπορεί να το κρίνει, γιατί σε τελική ανάλυση η απόφαση θα ληφθεί από την Ισλανδία. Ευχαριστώ εκπρόσωπος της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει το λόγο ο κύριος Χάνεκεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Εξωτερικών και τον Πρόεδρο για την πρόσκληση ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πράγματι θεμελιώδης όσον αφορά τα δημοκρατικά διαπιστευτήρια της διαδικασίας διεύρυνσης ακριβώς όπως βεβαίως ε, και η διαδικασία στο δικό μας κοινοβούλιο. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την εκτίμησή μου για τις τρεις ε, παρεμβάσεις που ακούστηκαν μέχρι στιγμής. και σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ με αυτή την ανάλυση. Να συνοψίσω εδώ πέρα το πού βρισκόμαστε εμείς η κυβέρνησή μας αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει. Η Ισλανδία όπως ξέρετε υπέβαλε αίτηση ένταξης 17 Ιουλίου 2009 27 Ιουλίου 2010 ξεκίνησαν επισήμως οι διαπραγματεύσεις και τώρα έχουμε την διαδικασία προενταξιακής εξέτασης. Αυτό σημαίνει βεβαίως το κεκτημένο το οποίο εξηγείται κεφάλαιο προς κεφάλαιο και εμείς εξηγούμε το τι κάνουμε στην Ισλανδία. Ελπίζω λοιπόν να συμφωνήσουν και οι συνάλφοι των την πως είναι σταθερός ο ρυθμός Εκτιμούμε την εξαιρετική συνεργασία με την ε, Κομισιόν και γνωρίζουμε το ότι υποφελούμαστε σε σύστημα συστήματο, συστήματος το οποίο είναι πολύ οργανωμένο και είναι μια διαδικασία βέβαιως ε, αυτή η ενταξιακή η οποία λειτουργεί καλά. Επίσης το μικρό μέγεθος της διοίκησής μας ε, κάποια από τα Υπουργεία μας έχουν το μέγεθος διευθύνσεων σε άλλες χώρες, αλλά παρόλα αυτά έχουμε πολλούς ειδικού και βεβαίως αυτή είναι η ειδική με 16 χρόνια εμπειρία στο να εφαρμόζουν την νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς και έρχομαι έτσι άρα στο δεύτερο σημαντικό θέμα γιατί όπως ξέρετε η Ισλανδία ήδη βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες. Ο συνάδελφος από την Κομισιόν ήδη ανέφερε τη συμφωνία ΕΟΧ. Υπάρχει σύνδεση με χώρος Σέγγεν, δικαιοσύνη και εσωτερικά, αλλά βεβαίως όπως αναφέρθηκε υπάρχει το γεγονός ότι ευθυγραμμιζόμαστε με όλες σχεδόν τις δηλώσεις ε, της ΚΕΠΑ. Επίσης προσφέρουμε μια πολιτική συμφωνία με την Ένωση για να εφαρμόσουμε περιορισμούς ε, στις εκπομπές ε, μόλις βεβαίως επιτευχθεί η διεθνής συμφωνία για την κλιματική πολιτική και έχουμε δηλώσει πως ε, θα συνταχθούμε με τους πιο φιλόδοξους ε, στόχους. Επίσης, ε, έτσι Δευτερευόντω, νομίζω πω είμαστε κάπω ασυνήθιστη υποψήφια χώρα με την έννοια πω έχουμε συνεισφέρει πολλά εκατομμύρια ευρώ ε, στη μείωση των ε, κοινωνικών ανισοτήτων στην Ένωση, επί σειρά ετών. επίση αναφέρθηκε πω θα έχουμε βέβαια κάποια δύσκολα κεφάλαια. Τα κεφάλαια αυτά έχουν ήδη αναφερθεί από τους συναδέλφους. Εγώ συμφωνώ οπωσδήποτε πως η αλληλεία είναι στο επίκεντρο. Περιφερειακή πολιτική, νομισματική πολιτική οπωσδήποτε. Αν και οι δυσκολίες τους δεν θα είναι τόσο μεγάλες, τόσο πολύ πολιτικές όσο τεχνικές. Αλλά ειδικά στη Γεωργία που είναι ένας τομέας κλειδί και στην Αλληλεία Νομίζω πως θα μας καθοδηγήσει εδώ πέρα το κοινοβούλιο μας και η σχετική του γνωμοδότηση του 2009 που καθόρισε το πλαίσιο εντός του οποίου θα διαπραγματευτούμε. Αν μου επιτρέπετε τώρα για αυτά τα οποία ακούστηκαν ο Άλτουρ Φόρατσον πολύ σωστά παρουσίασε τα πράγματα. Είπατε πως μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτου ε, σε μια δημοσκόπηση 63% του πληθυσμού ήθελε να συνεχιστεί η ενταξιακή διαδικασία. Δηλωμένος στόχος της κυβέρνησης είναι βεβαίως να υπάρχει μια διαφανής ε, τέτοια διαδικασία με ισορροπημένη πληροφόρηση του κοινού και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαίως τόνισε την σημασία του να ενημερωθεί σωστά το κοινό. Το γνωρίζουμε αυτό. Το δε κοινοβούλιο μας είναι εδώ πέρα, παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και η διοίκηση θα εργαστεί υπό τον έλεγχο του κοινοβουλίου. Αλλά για να σας δώσω μια ιδέα για το τι γίνεται ο επικεφαλής διαπραγματευτής και η ομάδα του έχουν ήδη ταξιδέψει τους μεγαλύτερους οικισμούς της Ισλανδίας και θα συνεχίσουν να το κάνουν, να εξηγούν, να αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες του κόσμου. Επιπροσθέτως έχουμε τώρα ένα διαδραστικό site όπου οποιοδήποτε μέλος του κοινού μπορεί να στείλει σχόλιο η ερώτηση σε οποιοδήποτε από τα κεφάλαια αυτά και να λάβει γρήγορα μια ουσιαστική απάντηση. Και ελπίζουμε με τον τρόπο αυτόν μαζί με ένα ευρύτερο διαπραγματευτικό πλαίσιο να ενημερωθεί το κοινό για την ουσία των διαπραγματεύσεων αλλά και για το τι σημαίνει η ένταξη στην Ένωση. και θα προσπαθήσουμε βεβαίω τις διάφορες ιδέες που υπάρχουν να τις μετατρέψουμε. Να τονίσουμε ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα να μην έχουμε έτσι μόνο αφηρημένες ιδέες. Υπάρχει βεβαίω, όπω ξέρετε, και η μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή Ένωση Ισλανδία, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό σε συμβολικό και σε ουσιαστικό επίπεδο. Και βεβαίω έτσι εμβαθύνονται οι διπλωματικέ σχέσει μεταξύ των δύο πλευρών. Πού πάμε από εδώ και μπρο. Η διαδικασία εξέταση νομοθεσία θα τελειώσει τον Ιούνιο. Ελπίζουμε λοιπόν να ανοίξουμε κάποια κεφάλαια. Από την άλλη, βέβαια, η διαδικασία πρέπει να έχει τη δική τη δυναμική, δεν είναι αγώνα δρόμου. Ε, και ελπίζουμε βέβαια να προχωρήσουμε ανάλογα με την ουσία των πραγμάτων. Για να τελειώσουμε. συνάδελφος ανέφερε το ζήτημα της Κουμπριού. Πράγματι η Ισλανδία είναι ένα από τα τέσσερα παράκτια κράτη και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να το λύσει αυτό, αλλά πρέπει να θυμάστε πως υπάρχουν τέσσερα, όπως είπα, τέτοια κράτη και είναι ευθύνη και των τεσσάρων να βρουν μια συμφωνία. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Οπότε δεν νομίζω να επηρεάσει καθόλου τη διαδικασία ένταξη. Είναι κάτι που αφορά το εξειδικευμένο αυτό φόρουμ. Τέλο, ε, επειδή αναφέρθηκε από πολλού, η Ισλανδία έχει τις δυνάμει εκείνες, ε, τι ε, πολιτισμικές, δημοκρατικές και πολιτικές που απαιτούνται και αυτό το έκρινε και η Κομισιόν και όπως είπε και η Υπουργός των Εξωτερικών μας στην πρώτη διάσκεψη το να βρούμε κάποιο κοινό τόπο μεταξύ των συμφερόντων της Ισλανδίας και των κοινών συμφερόντων της Ένωσης θα είναι βεβαίως μια πρόκληση που απαιτεί προσπάθεια και δημιουργικότητα και βεβαίως αναμένουμε με αισιοδοξία αυτή την πρόκληση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μετά τι παρεμβάσει των, ε, των φιλοξενωμένων δίνω το λόγο στον ε, εισηγητή. Α, ζητώ συγγνώμη. Ο κ. Γκραμ Avery έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Βιαζόμουν. Ζητώ συγγνώμη. Έχει το λόγο κύριε Avery. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι άλλοι ομιλητέ κάλυψαν όλα τα βασικά θέματα πλήρω και καλά. Τι να προσθέσω εγώ. Έχω μακρά εμπειρία με διευρύνσει. Πάνω από 40 χρόνια παλιά ήμουν ένα νέο μέλο τη βρετανική ομάδα που διαπραγματευόταν ε, την προσχώρηση τη Βρετανία και ήμουν ανάμεσα στου αρχιτέκτονε άλλων διευρύνσεων που ήμουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα είμαι στην κοινότητα προβληματισμού και ενδιαφέρομαι για την Ισλανδία. Αυτό μπορώ να κάνω εντό του πενταλέπτου που μου έχει διατεθεί είναι να θέσω το θέμα αυτό τη προσχώρησης της Ισλανδία σε ευρύτερο πλαίσιο και α πούμε και ιστορικό πλαίσιο και θέλω να πω τρία πράγματα εν συντομία. Πρώτα απ' όλα αυτή η διαδικασία της διευρύνσεως βασικά οδηγείται από τις υποψήφιες χώρες. Γιατί έχουμε την πολιτική διευρύνσεως επειδή οι ευρωπαϊκές γειτονικές χώρες χτυπούν την πόρτα και θέλουν να μπουν. We Εμείς στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ποτέ δεν θέλουμε τον κόσμο μας να ψάχνει και δεν ζητήσαμε την Ισλανδία να προσχωρήσει. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ζήτησαν, έκαναν έτοιμα ως Δική της ήταν η πρωτοβουλία όμως. Αυτό τι συνεπάγεται. Συνεπάγεται νομίζω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε δικαίωμα να περιμένουμε την Ευρωπαϊκή, από την Ισλανδία να αποδεχτεί τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κεκτημένο, τους στόχους της Ένωσης και αυτό ισχύει για τα πάντα. Αλληλεία, γεωργία, όπου εκεί βεβαίω μπορούμε να έχουμε ειδικέ διευθετήσει όσον αφορά την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων τη Ισλανδία, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε σε αυτού του τομεί αυτοεξαιρέσει. Εφόσον αναφέρθηκα σε αυτοεξαιρέσει, να προσθέσω ότι κάποια από τα κράτη-μέλη μα παραμένουν εκτό του Σέγγεν και του ευρώ. Αλλά η Ισλανδία είναι ήδη εντό ε, τη Σέγγεν και θέλει να ενταχθεί και στο ευρώ άλλη συνεπαγωγή της πολιτικής διεύρυνσης και επειδή είναι και πρωτοβουλία της Ισλανδίας είναι ότι οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας αυτής που ζήτησαν την ένταξη έχουν δικαιώματα και ευθύνε. Η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της κατά τις διαπραγματεύσεις της ένταξης. Θα το κάνει αυτό με θέρμη, αλλά έχει και την ευθύνη να εξηγήσει στον πληθυσμό της χώρας τους λόγους για τους οποίους η ένταξη είναι προς όφελος στρατηγικών συμφερόντων της ε, Ισλανδίας. Αν είναι επιτυχή τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων προσωπικά, εκφράζω την ελπίδα ότι στο δημοψήφισμα πετύχουν θετική απάντηση και θα ακολουθήσουν ε, τη διαδρομή της Νορβηγίας που πέταξε την κοιλάδα των λιγμών για να καταλήξει για την έγκριση της συνθήκης ένταξης και ο λαός είπε όχι. Ένας από τους λόγους που είπαν όχι οι Νορβηγοί ήταν και το πρόβλημα της αλίας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Κάτι άλλο θέλω να πω κύριε Πρόεδρε ότι η Ισλανδία είναι αρκετά διαφορετική από άλλες υποψηφίες χώρες. Διαφέρει από τις άλλες χώρες που είναι ήδη υποψηφία εντάξει, Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία και διαφέρει και από άλλη υποψήφια χώρα του παρελθόντος, ακόμα και από τις σκανδιναβικές χώρες που ήδη έχουν προσχωρήσει. Να αναφέρω ότι η Ισλανδία είναι η μικρότερη χώρα που υπέβαλε ποτέ υποψηφιότητα προσχωρήσεως, 320.000 πληθυσμό, εντελώ διαφορετική από την Τουρκία. Θα ήταν το μικρότερο κράτος μέλος. Είναι η πλουσιότερη χώρα που έκανε ποτέ αίτηση για προσχώρηση, πριν την οικονομική κατάρρευση είχε το υψηλότερο κατακεφαλήνα ΕΠ στην Ευρώπη και ακόμα το κατακεφαλήνα ΕΠ είναι πολύ ψηλό και είναι η καλύτερα προετοιμασμένη ψηφιακή χώρα που είχαμε ποτέ διότι ήταν στον ΕΟΧ για 16 χρόνια. Τώρα αυτή η διαφορά σημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε σοβαρά την αρχή της διαφοροποίησης. Η αρχή της διαφοροποίησης είναι θεμελιώδης για την πολιτική της διεύρυνσης και τι σημαίνει σημαίνει ότι εφαρμόζουμε τις ίδιες αρχές σε όλες τις υποψήφιες χώρες, αλλά λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητε της Ισλανδίας. Να δώσω ένα παράδειγμα. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι η Ισλανδία έχει το διοικητικό δυναμικό να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη Γεωργία και όλα τα άλλα. Ήδη εφαρμόζει το μισό κεκτημένο. Οπότε δεν χρειάζεται να εφαρμόσουμε τις ίδιες δοκιμές αντοχής στην Ισλανδία όπως κάνουμε στις αλγανικές χώρες. Και το τελευταίο σημείο, το τρίτο μου που έχω να τονίσω, είναι ότι η Ισλανδία δεν είναι μόνο διαφορετική αλλά και απόμακρη και δεν την καταλαβαίνουν πολύ καλά στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Καλύτερα να την καταλαβαίνετε εσείς εδώ στις αιθούσεις, εντός αιθούσεις από ό,τι άλλοι απ' έξω. Είναι περίπλοκη, δύσκολη χώρα να κατανοηθεί, έχει πολλά παράδοξα, είναι πολύ νεοκράτος, ήταν τελευταίο έδαφος που κατέκτησαν οι Βίκινγκς, που, που κατοικήθηκε από τους Βίκινγκς. Έχει το παλιότερο κοινοβούλιο όμως και την ε, πιο ε, παλιά λογοτεχνία στην ε, Ευρώπη. Είναι πολύ ιδιαίτερη χώρα. Δεν ξέρουμε αν θα πει ναι η Ισλανδία για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ιστορικέ και πολιτικέ συνεπαγωγέ αρνητική ψήφου ή θετική ψήφου μπορεί να είναι πολύ σημαντικέ, αλλά παρόλα αυτά η Ισλανδία μπορεί να επιβιώσει και, και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πει όχι η Ισλανδία, δεν θα κάνει τη μεγάλη διαφορά όσον αφορά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ή την ευρωπαϊκή ιστορία. Όμω παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα ήταν ντροπή οπισθοχώρηση ένα χαστούκι αν μια μικρή πολιτισμένη χώρα μας απορρίψει και γι' αυτό νομίζω ότι χωρίς να κάνουμε παραχωρήσεις επί των αρχών στις διαπραγματεύσεις με τη Ισλανδία για την ένταξη θα πρέπει να είμαστε επικοδομητικοί και πλήρη στην προσέγγιση να βοηθήσουμε τους Ισλανδούς να πετύχουν τελικά ένα νέο ναι από το λαό της Ισλανδίας. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά θέλουμε την άποψη του εισηγητού του συναδέλφου του κ. Πρέντα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά τους προσκεκλημένους μας που είχαν την καλοσύνη να έρθουν στο σημερινό σεμινάριο και να μας κάνουν τις παρουσιάσεις τους που ήταν όλες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αλλά και πολύ χρήσιμες και θα αποφανούν χρήσιμε και για την έκθεση που καταρτίζω για την ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Είμαι ο για την Ισλανδία και την ένταξη της Ισλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά πάσα πιθανότητα θα συζητήσουμε αυτή την έκθεση το Φεβρουάριο το Μάρτιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευελπιστούμε ότι θα περάσει αυτή η έκθεση στην Ολομέλεια του Απριλίου στο Στρασβούργο. Με την άδειά σας θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για τα θέματα που ακούσαμε και να υποβάλω και ορισμένες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Θόρκαρσον για τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε την θέση της Ισλανδίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν πολύ εξειδερκής οι παρατηρήσεις του και είπε ότι όπως εντάχθηκε η Ισλανδία στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο έχουμε ουσιαστικά τους σοσιαλδημοκράτες μόνο ένα κόμμα που είναι αναφανόν υπέρ της ένταξης της Ισλανδίας. Θα δούμε αν στεφθεί με επιτυχία ε, το σχέδιο αυτό και η προοπτική αυτή και μετά την ένταξη στον ΕΟΧ, παρόλο που δεν τη χάνει γενικότερη υποστήριξη αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπέιλς, γιατί μας παρουσίασε τη στρατηγική θέση της Ισλανδίας, σε μια στιγμή μάλιστα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαμορφώσει τη θέση της και ως προς την αρκτική ζώνη. θα εξετάσουμε και την έκθεση Γκάλερ για τον απότερο βορρά. Είναι επίκαιρο λοιπόν το θέμα και της αρκτικής ζώνης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Ντέιβιτ Κέρι για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή του ως προς τα οικονομικά και τα δημοσιονομικά ζητήματα. Εκεί ε, μας ανέλησε τα υπέρ και τα κατά για την Ισλανδία, αλλά μας ανέλησε και τον συμβολικό και συγκινησιακό χαρακτήρα της ενδεχόμενης ένταξης της Ισλανδίας. Θα ήθελα να υποβάλω τρεις ερωτήσεις στους προσκεκλημένους μας. Καταρχήν μια ερώτηση προς την κυρία Μπέιλς. Θα ήθελα να μιλήσω για τις θετικές σχέσεις που έχει η Ισλανδία με τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά προτιμώ να επικεντρωθώ στις σχέσεις της Ισλανδίας με τη Ρωσία και να Αναφερθώ και στην πρόταση του κυρίου Γκράχαμ Έιβορη για τις πρόσφατες διευρύνσεις. Η πλειοψηφία των ε, κρατών μελών εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν μέσω τεταμένων σχέσεων με τη Ρωσία εξαιτία του σοβιετικού του παρελθόντος. Στην περίπτωση της Ισλανδίας έχουμε μια διάσουσα περίπτωση αγαστών σχέσεων με τη Ρωσία. Διαρωτώ με λοιπόν, συμφέρει τη Ρωσία μία ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ρωτώ αυτό στα πλαίσια και τη συζήτηση για τον απότερο βορρά. Τι θα κερδίσει η Ρωσία από μια ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα κερδίσει ως προς τη θέση της στον Αρκτικό Βορρά. Η δεύτερη μου ερώτηση απευθύνεται στον κύριο Τόρχαλσον. Τη Δευτέρα η Ισλανδική Βουλή θα λάβει θέση ως προς τη νέα συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο και την, Ολλανδία, και την ε, Ολλανδία για το ΆΙΣΕΒ, για τη διάσωση του πάγου. Ποια είναι τα πιθανά σενάρια. Αν η Ισλανδική Βουλή υπερψηφίσει αυτή τη συμφωνία με την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η δημόσια συζήτηση στην Ισλανδία θα επικεντρωθεί περισσότερο στο, στο θέμα της ένταξης ή αν απορριφθεί αυτή η συμφωνία. Πιστεύετε ότι η Ισλανδική κοινή γνώμη θα στραφεί και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά της ένταξης Ευρωπαϊκής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Κέρι αναφέρθηκε στο συμβολικό και συγκινησιακό χαρακτήρα αυτής της Απόφαση ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς λοιπόν πιστεύετε κύριε Κέρι ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη συζήτηση στην Ισλανδία γιατί κάποια κόμματα που τάσσονται υπέρ της ένταξης προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε ευκαιρία συζήτηση και οποιαδήποτε δήλωση που γίνεται για την Ισλανδία ως απόδειξη, ως περίτρανη απόδειξη της ανάμειξης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα Ισλανδικά ζητήματα. Αυτά είναι επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι πολέμοι της ένταξης. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Ισλανδία για να έχει μια ισορροπημένη συζήτηση για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. η Μήπω η παρουσία οποιοδήποτε εκπροσώπου τη Ένωση μπορεί να εκλειφθεί ω παρέμβαση τη Ένωση στα εσωτερικά πράγματα. Λοιπόν, θα μαζέψουμε και τι ερωτήσει και των άλλων συναδέλφων θέλουν να παρέμβουν. Ο καθένα έχει στη διάθεσή του δύο λεπτά. Κυρία Γκόμες, Κορνέλισεν, Φέρμ και Τάνοκ είναι οι συνάδελφοι να μιλήσουν. Κυρία Γκόμες, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, παρουσιάσεις. Εγώ είμαι από, την άλλη άκρη της Ευρώπης, την Νότια Πορτογαλία. Και προβληματίζομαι αλλά και ικανοποιούμε από την άλλη που πραγματικά συζητούμε την προσχώρηση της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβληματίζομαι γιατί. Εντάξει, καταλαβαίνω το λόγο, λόγω της κρίσης, οικονομικής κρίσης. Η Ισλανδία, η Ισλανδοί μάλλον αισθάνθηκαν ότι είναι ασφαλέστεροι μπαίνοντας στην κρίσιμη μάζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. E Αλλά αναρωτιέμαι διότι κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποια κράτη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυσαρεστημένα όσον αφορά το πώ λειτουργήσε, όσον αφορά το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συζητείτε. Συζητούν κάποιοι να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι δική μου άποψη. Εξεπλάγει όταν το 2008-2009 θαρώ συμμετείχα στην κοινοβουλευτική συνέλευση συνελεύσεις του ΝΑΤΟ και είδα τους διπλωμάτες, τους συναδέλφους ε, της Ισλανδίας και τους βουλευτές που είχαν εξοργιστεί κατά των μέτρων που είχαν εφαρμοστεί ε, επί της Ισλανδίας από Ολλανδία, Βρετανία λοιπά Τους αντιμετώπισαν σαν τρομοκράτες λόγω της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης που πέρναγε η Ισλανδία. Και εγώ έδειχνα μεγάλη κατανόηση, τους καταλάβαινα τους Ισλανδούς. Βέβαια, ούσα Πορτογαλίδα έχω ιδιαίτερου δεσμού με την Ισλανδία. Γιατί εμεί τρώμε μανιωδώ τον μπακαλιάρο τη Ισλανδία. Άρα έχουμε ισχυρού δεσμού που χρονολογούνται από παλιά, εδώ και πολλούς αιώνες που συνεργαζόμαστε στην αλία του μπακαλιάρου. Άρα, από τη δική μου εμπειρία πρέπει να πω ότι οι Ισλανδοί είναι σκληροί διαπραγματευτές. Προστατεύουν τα συμφέροντά τους. Θα προστατεύσουν την αλληλεία τους και τη γεωργία τους στις διαπραγματεύσει. Και αυτό ίσω να μην είναι πρόσδεκτο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σίγουρα είναι μια συνταγή για ένα καλό μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αν γίνει μέλος η Ισλανδία θα είναι ικανοποιημένη, θα θέλει να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχυρό προσπιστή τη Ισλανδία, κύριε κυρία Γκόμε, λέει ο πρόεδρο. Η κυρία Κορνέλησαν τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους για τις πολύ ενδιαφέρουσε ε, παρουσιάσεις σας. Έμαθα ξανά πολλά. Ερώτημα για την αλία. Πολλοί από εσά τονίσατε ότι αυτό θα είναι ένα από τα ακανθόδη από τα δύσκολα αποφασιστικά θέματα όσον αφορά την προσχώρηση της Ισλανδίας. Θέλει συμφωνία, χρειάζεται συμφωνία από αυτού η Ισλανδία. Ο κύριος Avery, Avery είπε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει opt-out αυτοεξαίρεση. Εγώ θα έλεγα βλέποντας την ανωτερότητα της αλληλευτικής πολιτικής της Ισλανδίας δεν θα ήταν κακή ιδέα μια αυτοεξαίρεση Ισλανδίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Σκάρη μπορούν να μου απαντήσουν σε κάτι. Ποιε είναι οι επιλογές. Ένα opt-out ε, είναι επιλογή. Τι άλλες επιλογές υπάρχουν. ούτω ώστε η Ισλανδική αλληλευτική πολιτική να παραμείνει ακέραια σε τέτοιο βαθμό, ούτω ώστε να εξακολουθεί να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της Ισλανδία. Κύριος Φέρμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι πραγματικό μέλο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ο οποίο μέλο τη Επιτροπή Προπολογισμών και συγγετή για τη διεύρυνση στην Ελόγω Επιτροπή. Είμαι Σουηδό Σοσιαλδημοκράτη, να καταλαβαίνω κάποια από τα σκανδιναβικά χαρακτηριστικά τη χώρα και υποστηρίζω και την ε, προσέγγιση του Δημοκρατικού Κόμματο, του Αδελφού Κόμματο στην Ισλανδία, που είναι υπέρ τη Ευρώπη. Σε αυτά που είπε η κυρία Κορνέλη, να συνεχίσω κι εγώ. Η Αλία και η Γεωργία και κάποιοι άλλοι τομεί, όπω γνωρίζουμε, ίσω να είναι προβληματικοί τομεί για τι διαπραγματεύσει. Το ερώτημά μου είναι πιο συγκεκριμένο όμω. Ήδη ε, υπάρχει απόφαση στην Ισλανδική κυβέρνηση, στο Κοινοβούλιο τη Ισλανδία, όσον αφορά τα αιτήματα για συγκεκριμένα opt-outs. Υπάρχουν τομεί συγκεκριμένοι όπου θέλετε εξαιρέσει από το κεκτημένο Ευρωπαϊκή Ενώση, μεταβατικού κανόνε, οτιδήποτε μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένο και είναι ένα ερώτημα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που ευθύνω τώρα. Τώρα ήδη βλέπουμε που έγκυνται τα προβλήματα των διαπραγματεύσεων. Πιο συγκεκριμένα, εκτό από γενικόλογα να λέμε αλλιευτική πολιτική, πού θα θέλατε δυνατότητες εξαιρέσεων, αυτοεξαιρέσεων, opt-outs. Ο συνάδελφό μα, ο κύριος Τάνοκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας αυτή και το πάνελ και τους διακεκριμένους ε, προσκεκλημένους μας και ειδικά τα όσα ακούστηκαν από τον Κρέα Μέιβερη. Εγώ, ξέρετε, η χώρα μου έχει το Ηνωμένο Βασίλειο στενούς ιστορικούς ε, δεσμούς ε, με την Ισλανδία. Στην Οξφόρδη όταν σπούδασα ιατρική είχαμε πολλούς Ισλανδούς συμφοιτητές γιατί δεν είχαν ιατρική σχολή στο Ρέικιαβικ. Και βεβαίως είχαμε και τον πόλεμο του Μπακαλιάρου τη δεκαετία του 70, αλλά έχει περάσει καιρός από τότε. Εγώ θα ήθελα βεβαίως να πούν ναι στο δημοψήφισμα, αλλά θα είναι τσίμα τσίμα τα πράγματα και θα είναι παρόμοια η κατάσταση με τη Μάλτα, ένα άλλο μικρό κράτος μέλος που είχε πολλωμένη κοινή γνώμη όσον αφορά την ένταξη, αλλά τα πράγματα έχουν έκτοτε επιληθεί. Οπωσδήποτε, καθώς προέρχομαι από το, το κόμμα στο οποίο προέρχομαι, πιστεύω στην κοινή αλληλευτική πολιτική και θεωρώ και ελπίζω η διαδικασία ένταξης της Ισλανδίας να καταλήξει σε μεγάλες παρεκκλήσεις ε, αν όχι και σε προσπάθειες μεταρρύθμισης της κοινής αληφτικής πολιτικής γιατί βεβαίως έχει χρεοκοπήσει εδώ και χρόνια αλλά ελπίζουμε έτσι να ενταχθεί και η Νορβηγία κάποτε στο μέλλον εάν διασφαλίσουμε πως η αλληλεία δεν αποτελεί εμπόδιο σε χώρες σαν την Νορβηγία τις οποίες επίσης θα θέλαμε να καλωσορίσουμε στο μέλλον. Είμαι και ο για την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών. Οπωσδήποτε υποστηρίζουμε την ένταξη της Ισλανδίας και το Μαυροβούνιο την άλλη πολύ μικρή υποψήφια χώρα που επίσης ε, και αυτή βεβαίως είναι στα ωριά της όσον αφορά τις διοικητικέ δυνατότητες της και δεν είναι καν μέρος του, μέλος του ΕΟΧ. Χαίρομαι που ακούω πως το πρόβλημα με τη τράπεζα iSave μάλλον έχει επιληθεί πλήρως ως αποτέλεσμα των χαμηλών επιτοκίων που έχουν συμφωνηθεί για την αποπληρωμή του χρέους. Επίσης συμφωνώ πως υπάρχει πρόβλημα με την υπεραλληλία του σκουμπριού. Αυτό το οποίο με ενοχλεί είναι όταν βγαίνει η Κομισιόν και δηλώνει διάφορα κατηγορηματικά πράγματα. Δεν ξέρω με τι νομική βάση και μιλάει για την αλληλεία φαλενών μink ε, μικρής κλίμακας που γίνεται και λέει πώ έτσι παραβιάζεται το κεκτημένο. Κατά την άποψή μου νομίζω πως είναι κοινή θέση όλων των ε, κρατών μελών στην ΚΕΠΑ το μορατόριο στη Διεθνή Επιτροπή φαλαινοθύρια. Αλλά το να λέμε τώρα παραβίαση του κεκτημένου, ποια νομοθεσία παραβιάζεται. Δεν σημαίνει πως όλες οι κοινέ θέσει εξωτερική πολιτική είναι δεσμευτικέ για εξωτερικέ χώρε. πριν ενταχθούν. Επίσης, Δεν ξέρω, μίλησε ο κύριος Πρέντα για πολυπολική εξωτερική πολιτική της Ισλανδίας. Δεν ξέρω, νομίζω πως ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ έχουν μια συγκεκριμένη πολιτική. Εντάξει, έχουν σχέσεις με την ε, Ρωσία, δεν το ήξερα αυτό, αλλά ελπίζω αυτό να μην παίζει ρόλο στη διαδικασία ένταξης. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ωραία, δεν ζητά άλλο το λόγο. Άρα, στα μέλη του πάνελ αναθέτω να απαντήσουν στις ερωτήσεις που ετέθησαν τους συναδέλφους. Ο καθένας σας έχετε δύο λεπτά και αποφασίστε ποιος θα μιλήσει πρώτος και σε ποιες ερωτήσεις θα απαντήσει. Ενώ παίρνετε εσείς τη δύσκολη απόφαση να πω στους συναδέλφους εγώ ότι το σχέδιο ψηφίσματος του κυρίου Πρέντα για την Ισλανδία θα εξεταστεί για σύντομη ανταλλαγή απόψεων, πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή ΑΦΕΤ στις 10 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους και δίνω το λόγο σε όποιον θέλει να, να μιλήσει, να δώσει απαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ενδιαφέρουσα ερώτηση για τη Ρωσία. Ε, ούτε και στο, στη σκανδιναβική περιοχή δεν είναι ιδιάζουσα η θέση της Ισλανδίας και η Δανία δεν θεωρεί κίνδυνο τη Ρωσία, αλλά και η ε, Νορβηγία υποτιθέλει θετική συνεργασία με τη Ρωσία και αυτό αναφέρεται στη φαλαινοθυρία και σε κοινή ε, θαλάσσια διαχείριση. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα η Ισλανδία διοργάνωσε μία ε, συνεδρίαση στην οποία συμμετείχε και η Ρωσία για την κοινή έρευνα και διάσωση διάσωση, κάτι που είναι σημαντικό επίτευγμα. Άλλωστε και η Ρωσία με την ένταξη θα έχει μια θετική δανεία παρόμοια με αυτή που ασκείται εκ μέρους της δανείας για την Γρυλανδία και, και την Ορβηγία που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, η Ισλανδία, μετά την απόσυρση των ε, Αμερικανικών βάσεων και την οικονομική κατάρρευση η Ισλανδία μπήκε στον πειρασμό να ψάξει νέου φίλους και μάλιστα είχε την ψευδέση ότι θα λάβει ε, δάνειο από τη Ρωσία κάτι που τελικά δεν επιβεβαιώθηκε. Νομίζω ότι ευελπιστώ ότι θα απομακρυνθεί δηλαδή, από τη Ρωσία από τη στιγμή που θα λάβει τη στρατηγική υποστήριξη με την ε, ένταξη ενδεχομένω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και συγγνώμη για τη σύντομη απάντηση. Ό,τι αφορά το iSave. Βέβαια, ένας ε, επιστήμονας ε, πολιτικών επιστημών δεν επιχειρεί προγνωστικά για το μέλλον. Εγώ πιστεύω πάντως ότι μάλλον το, το, η Βουλή θα εγκρίνει τη συμφωνία και ίσως όπως και στο παρελθόν θα παραμένει στο θέμα σε δημοψήφισμα. Βέβαια και πάλι υπάρχει πιθανότητα να καταψηφίσουν οι ψηφοφόροι αυτό το θέμα. Μετά θα αποφασίσει ο πρόεδρος. Πάντως, αν η Ισλανδική Βουλή δεχθεί την συμφωνία για το ISF και προσυπογράψει το διάταγμα ο πρόεδρος, μπορούμε για μια διετία να βγάλουμε το κεφάλι μας σε αυτό το θέμα και να επικεντρωθούμε στο θέμα της ένταξης. Σε ό,τι αφορά την αλία, είναι σημαντικό να ε, επισημάνουμε ότι ένα τμήμα μόνο της Ευρώπης, της βόρειο-δυτικής Ευρώπης ε, που ε, δεν ενδιαφέρεται για αυτό το σχέδιο. Εδώ μιλούμε για κράτη. Τη όπως η, Νορβηγία, η Ισλανδία, οι νησίες Φερόες, η, η Γρυλανδία που έχουν αυτή την απροθυμία εξαιτία της αλήθειας κυρίως. Είναι τέσσερις χώρες που δεν ενδιαφέρονται τόσο να στραφούν προς την Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να φτάσει προς αυτές για την Αλία. Η Ισλανδία διεκδικεί την ε, ε, διεκδικεί την δυνατότητα να διαχειρίζεται από μόνη της την αλληλεία της, κάτι που έχει επιτυχώς πραγματοποιήσει όλα τα χρόνια μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω λίγο στους τελευταίους που ρώτησαν για τα opt-out. Βεβαίως, είναι ζήτημα αρχής να μην ε, δίνουμε opt-out ε, στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Ε, είναι πολιτικό γεγονός. Εάν επιτρέπαμε στα νέα μέλη να έχουν τα ωφέλη χωρίς υποχρεώσεις της ένταξης, τι θα γινόταν και τα παλαιά μέλη θα ζητούσαν τα, ίδια προνόμια. Οπωσδήποτε πρώτοι οι Βρετανοί και μετά θα ακολουθούσαν όλοι οι Οπότε είναι ζήτημα αρχή στι ενταξιακέ διαπραγματεύσει. Να αποφεύγουμε την αποσταθεροποίηση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε να έχουμε κάποιες ειδικέ ρυθμίσεις. Παραδοσιακά η έξυπνη λύση ήταν μια μεγάλη μεταβατική περίοδος με ρήτρα αναθεώρησης. Και αυτό μου φαίνεται πως είναι η καλύτερη επιλογή στην ε, περίπτωση της αλληλείας. Πριν από δύο χρόνια η Κομισιόν έγραψε μια πράσινη βίβλο για την αλληλεία. Θα την είχατε διαβάσει, εγώ την έχω εδώ. Ένα ε, θαυμάσιο έγγραφο. Ξεκινά ο συγγραφέας με ένα όραμα για την Ευρωπαϊκή Αλληλεία το 2020. Να το να σας διαβάσω από μέσα. Μιλάει για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ε, πολιτική αλληλεία που θέλουμε στο μέλλον. Και λέει το 2020 η υπεραλία ανήκει στο παρελθόν, η κοινή πολιτική αλληλεία είναι απλούστερη και φτηνότερη. Δηλαδή όταν το διαβάζω λέω, ο, εδώ πέρα περιγράφεται η Ισλανδία. Ναι, πρέπει λοιπόν νομίζω να δούμε το ζήτημα της αλληλείας στο πλαίσιο του. Δεν είναι η Ισλανδία με χαμηλότερες προδιαγραφές από εμά. Γενικότερα, πλην εξαιρέσεων, έχει υψηλότερες προδιαγραφές. Δεν είναι ότι εν μία νυχτή θα πρέπει να προσαρμοστεί. Ευχαριστώ. Να πω ξανά αυτό που έλεγα την αλληλεία δεν είναι θέμα αυτοεξαίρεσης όταν λέει κοινή αληφτική πολιτική στα, θα αλλάξει. Δεν θα είναι αυτή που περιγράφει το έγγραφο του 2009. Θα κινηθεί προς την κατεύθυνση διαχειρίσεως των ε, αλλιευμάτων ε, με τον Ισλανδικό τρόπο. Ο Ισλανδός συνάδελφος μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό που λέω. Το Ισλανδικό Κοινοβούλιο έχει ένα έγγραφο στην σελίδα του και λέει τι ζητά από τι διαπραγματεύσει. Δεν το κατέβασα, άκουσα ότι υπάρχει όμως. Το άκουσα όταν ήμουν στην Ισλανδία ότι υπάρχει. Όσον ευρωπαϊκά, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και πώς επηρεάζουν τη συζήτηση, τις συζητήσεις. Δεν αφορά την παρεμβολή τρίτων. Η Ισλανδική κυβέρνηση συνεργάστηκε θετικά με το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ. Υιοθέτησε το πρόγραμμα, το στερνίστηκε Ισλανδία. Άρα όταν οι τρίτοι συνεργάζονται για κοινού στόχου με την Ισλανδία δεν υπάρχει πρόβλημα χορηγήσεων συμβουλών προς την Ισλανδία. Και θα πρέπει αυτοί που να έξω να δείξουν ότι καταλαβαίνουν τη θέση των Ισλανδών. Και πιο σημαντικό τομέα ζωτική σημασία είναι ο τομέα τη Αλία. Εκεί πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη αυτό και να ακολουθηθεί σωστή προσέγγιση. Ο κ. Χάνεγκεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συντομότατα, για δύο ερωτήσει. Πρώτον, αν πήραμε απόφαση επί συγκεκριμένων opt-outs. Ακόμα εξετάζουμε το θέμα. Οι διαπραγματευτικές μας ομάδες δεν έχουν ετοιμάσει ακόμα το διαπραγματευτικό πλαίσιο. Πολύ νωρίς να πούμε. Σε γενική αρχή όμως, από την άλλη πρέπει να πω δεχτήκαμε ότι παρεκκλήσεις, εξαιρέσεις δεν χρειάζονται εν γέννη. Πιστεύουμε και ιδιαίτερα στην αλληλεία ότι με δημιουργικότητα και ειδικέ ρυθμίσεις όπως ανέφερε ο κ. Σέιβερη μπορούμε να πετύχουμε αυτά που χρειαζόμαστε στο υφιστάμενο πλαίσιο. Σύντομα τώρα, στο θέμα των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, τη συζήτηση της ένταξης στην Ισλανδία. Ο πολιτική ζωή στην Ισλανδία είναι εξίσου πολύ, ε, περίπλοκη όπως και αλλού. Και σε ζωηρή δημοκρατική συζήτηση που συνεχίζεται ακόμα, είναι ξεκάθαρο ότι κάποια κόμματα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να υπονομεύσουν επιχειρήματα που δεν υπέρ τους. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι είναι σημαντικό να είναι ισορροπημένες οι πληροφορίες, αμερόληπτες πληροφορίες αυτές που δίνονται στο λαό, για να αποφασίσει έτοιμος πια ο λαός σε δύο-τρία χρόνια, όταν έρθει η στιγμή του δημοψηφίσματος. Αυτά και ευχαριστώ. Και για να κλείσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. To me. Uh, first... Uh, Καταρχήν, για την Αλία, αλλά και για οποιοδήποτε κεφάλαιο, εμείς διαπραγματευόμαστε το κοινοτικό κεκτημένο. Δηλαδή τα κράτη-μέλη διαπραγματεύονται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διαμεσολαβητή. Οι διαπραγματεύσει γίνονται μεταξύ των κρατών μελών και τη υποψήφια χώρα. Και αν τα κράτη-μέλη αποφασίσουν τι θα δώσουν και τι δεν θα δώσουν, ποιε παραχωρήσει θα κάνουν, ποιε υποχωρήσει θα κάνουν και θα ελέγχουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασία. Πάντω θα πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση. Δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί το κεκτημένο μέσω των διαπραγματεύσεων, μέσω των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Αυτή είναι η οροθετική γραμμή. Η αλλαγή του κοινοτικού κεκτημένου γίνεται σε, σε άλλο φόρουμ. Επίσης, ε, το ελευτικό κοινοτικό κεκτημένο είναι αυτό που αποτελεί τη βάση των διαπραγματεύσεων και στα πλαίσια τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Βέβαια, η Ισλανδία γνωρίζει ότι αυτό το κεκτημένο μπορεί να αλλάξει ανα πάσα στιγμή και παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ εξελίξει. Αν και όταν η Ισλανδία ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινοτικό κεκτημένο που θα εφαρμοστεί είναι το κοινοτικό κεκτημένο που ισχύει εκείνη τη στιγμή, τη στιγμή τη ένταξη. Και αυτό είναι σαφέ και ισχύει για οποιοδήποτε διαπραγματευτικό κεφάλαιο υπάρχουν σημαντικά θέματα για τις ρήτρες αυτοεξαίρεσης, τα opt-outs. Ε, οι ρήτρε αυτοεξαίρεση ε, συνιστούν ουσιαστικά αλλαγέ εκτιμένων που ισχύει για ορισμένε χώρε μέλη και που δεν εφαρμόζονται σε όλε. Εμεί είπαμε ότι, τα κράτη-μέλη δηλαδή, είπαν ότι δεν θέλουν να ισχύουν ε, δυνατότητες πλέον ρητρών αυτοεξαίρεση. Θέλουν να αποκλειστούν αυτέ οι ρήτρε αυτοεξαίρεση. Βέβαια, η Ισλανδία θα μα παρουσιάσει τη διαπραγματευτική τη θέση μετά το διεξοδικό έλεγχο, το screening. Εμείς ήδη έχουμε ελέγξει διεξοδικά, ολοκληρώσει το screening για 16 κεφάλαια. Θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία τον Ιούλιο και εκεί θα δούμε τις διαπραγματευτικές θέσεις και θα δούμε ποια είναι τα αιτήματα της ε, Ισλανδίας αν ε, υποβάλλει αίτημα αυτοεξαίρεση. Πάντως είναι καθησυχαστικά αυτά που μας είπε ο Νίκολας. Νομίζω ότι με το ισχυοκεκτημένο θα διευθετηθούν τα προβλήματα της Ισλανδίας. Σε ό,τι αφορά τη φαλαινοθυρία, ε, αντίκειται στο κοινοτικό κεκτημένο, το περιβαλλοντικό, όχι το αλλιευτικό. Γιατί για το περιβαλλοντικό κεκτημένο μιλάει για τη διαφύλαξη του οικοσυστήματος και των ε, διαφόρων αλλιευτικών ειδών. Και η φαλαινοθυρία αντιβαίνει σε αυτό το στόχο. Γιατί εμείς προσπαθούμε να διαφυλάξουμε ήδη ε, όπως της φάλαινας ε, ή κάποια άγρια πτηνά που θέλουμε επίσης να προφυλάξουμε. Αυτά είναι τμήματα του περιβαλλοντικού κοινοτικού κεκτημένου και σε αυτό αντιβαίνει η φαλαινοθυρία και νομίζω ότι ήδη αυτό το έχουμε τεκμηριώσει ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε λάβει και τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών και το αναφέρουμε και στην έκθεση προόδου. Δεν ξέρω αν υπήρχε άλλη ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι υπεράνω πάσης αμφιβολίας. Κύριε Διαδικαστικό, κύριε Τάνοκ. Όχι, απλώς ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Αναφερθήκατε στο θέμα της παλαινοθυρίας. Είπατε ότι εντάσσεται το κεφάλαιο το περιβαλλοντικό. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Σφάζονται οι φάλαινες και αλλιεύονται άλλα είδη ε, ε, φάλαινας που δεν κινδυνεύονται, δεν είναι στο κατεγραμμένες σαν κινδυνεύουσες, σαν κινδυνεύοντα είδη, όπως αυτά που κυνηγούν οι Ιαπωνέζοι. Δέχεται η Ισλανδική κυβέρνηση αυτή την προσέγγιση. Οι Δανείοι σχεδόν απομακρύθηκαν από τη συμφωνία, την κοινή θέση, ε, για την άρση του μορατόριου στην, ε, Πώ διαπραγματεύονται στην Επιτροπή για τη φαλαινοθυρία τη διεθνή, κάποια κράτη-μέλη και απ' την άλλη λένε ότι είναι κοινοτικό κεκτημένο η φαλαινοθυρία, η απαγόρευσή τη. Ο κύριο Χάναγκαν, πώ το ερμηνεύει το θέμα τη φαλαινοθυρία. Αυτό μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητο. Γιατί ίσω να παρεύουμε σε μακρά πρακτική που ακολουθείται στην Ισλανδία σε πολύ μικρή κλίμακα. Δεν ε, γίνεται υπεραλίες, δεν γίνεται μεγάλη αλία, μεγάλης κλίμακας των φαλενών και εξαγωγή του προϊόντος. Νομίζω ότι είναι πολύ ευαίσθητο θέμα εκεί και μπορεί να κολλήσουν οι διαπραγματεύσεις. Αυτή ήταν η ομιλία του κύριου Τάνοκ, η αγόρευση του κύριου Τάνοκ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Νομίζω πως θέσατε ένα σημαντικό ζήτημα και πράγματι το δάκλειο από των ήλων όταν είπατε πως είναι μια παραδοσιακή πρακτική από Ισλανδική σκοπιά βεβαίω έτσι είναι και είναι ενδιαφέρον πως η πράγματι είναι και εκτιμένο του περιβάλλοντος και είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζει το Υπουργείο Αλίας. Είναι ένας θαλάσσιος χώρος ε, εμείς ε, είμαστε υπέρ ε, της ε, αηφόρου εκμετάλλευσης θαλασσίων πόρων. Και αυτή εξακολουθεί να είναι η θέση μας και στην Επιτροπή Φαλονοφυρίας. Αλλά... Και... Μάλιστα. Να αναφέρω και την γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου μας, γιατί όπως σας είπα αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε διαπραγματευτική θέση, η θέση του Κοινοβουλίου μας λέει πως λέει πως ε, πρέπει να δούμε τι είναι η φόρο εκμετάλλευση ορισμένων ειδών στις διαπραγματεύσεις. Ε, πέραν τούτου δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ όλους. Αυτά ήταν όλα εμπειρογνώμονε συναδέλφου και κομισιόν. Η επόμενη συνεδρίαση 17 Ιανουαρίου. 7 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ.